We're going to start. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Εγκρίνεται. Περνάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη. Σα ενημερώνουμε ότι θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπή ε, στο Στρασβούργο τη Δευτέρα το βράδυ. Ε, η ημερομηνία δεν έχει ακόμη... Ε, τις 5 Εβδόμου, συγγνώμη, η ώρα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και το σχέδιο έκθεσης για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και το πλαίσιο σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην Ευρωζώνη. Δεύτερη ανακοίνωση. Σας ενημερώνουμε ότι η ακρόαση με τον Αλγίρδα Σέμετα που είναι ο Επίτροπος ε, για την ε, Φορολογία ε, και την Τελωνιακή Ένωση θα λάβει χώρα στις 3 η ώρα, στις 28 Ιουνίου, από τις 3 ως τις 4.30 στην ε, Γιάν 2Q2. Ε, Είναι τμήμα του διαρθρωτικού διαλόγου που η Επιτροπή μας ε, έχει σε τακτική βάση με τους Επιτρόπους για τομείς πολιτικής της αρμοδιότητός μας. Ναι, θα σας παρακαλούσα να επαναλάβετε το θέμα για το οποίο θα συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο Στρασβούργο. Σας είναι εύκολο. Δεν Θα παρακαλούσα να επαναληφθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο. Ναι, είναι η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα της Ευρωζώνης, στην Ευρωζώνη. Εντάξει. Θέλετε το λόγο? Όχι. Περνάμε στο σημείο 3 Τη ημερήσια διάταξη. την εξέταση των τροπολογιών. Κατευθυντήριες γραμμέ για τι πολιτικέ απασχόλησεις των κρατών μελών. Ο κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Εδώ πίσω είμαι. Στα αγγλικά ο κύριος Μάρτιν. Αρχίζω στα αγγλικά. Ε, χάρηκα πάρα πολύ και εκτίμησα πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε με τους συναδέλφους και τους βοηθούς και τη γραμματεία να συνεργαστούμε ε, γιατί ήταν πολύ πιεσμένος ο χρόνος και τελικά ε, ήμασταν και πολύ παραγωγικοί και πολύ αποτελεσματικοί. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι ήταν καταπληκτική αυτή η δουλειά και είμαι και πολύ ευγνώμων. Και περνάω στα γερμανικά τώρα. Εδώ μπορεί να φαίνεται ότι να μοιάζει επουσιώδες το θέμα, αλλά δεν είναι καθόλου επουσιώδες. Ε, αρκεί να δει κανείς και μόνο πόσες τροπολογίες έγιναν και με ποιες λεπτομέρειες από διάφορες πολιτικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κάθε ομάδα εδώ να δείξει ε, τι την ενδιαφέρει, να ανοίξει τα χαρτιά της. Έχουμε τροπολογίες κυρίως από τους αριστερούς, τους σοσιαλδημοκράτες και ε, τους συντηρητικούς αν είδατε τις απολογίες, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι ε, μεγαλύτερη σαφήνεια από αυτό που είναι πρόθυμο να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της για το 2020. Είχαμε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων, 16 ήταν οι δικές μου αρχικές τροπολογίες, έγινε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές και άλλους βουλευτές ε, ε, βοηθούς με πάρα πολύ ψηλά προσόντα και γνώσεις και τελικά τι αποκρισταλώθηκε ως βασική ιδέα. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιφύλαξη στην, ομάδα στην Επιτροπή μας συγγνώμη, να προχωρήσει στην επιλογή στόχων νέων και πιο ε, φιλόδοξων από αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύριο θα δείτε και στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, να υπάρχει η δυνατότητα για αυστηρότερους στόχους και αυστηρότερες ρυθμίσεις. Είτε πρόκειται για την απασχόληση των γυναικών και των ανδρών. Για παράδειγμα να πούμε τουλάχιστον 75% ανδρών και γυναικών και ε, πιο ηλικιωμένων Εγώ αγωνίστηκα για ένα στόχο και θέλω ακόμα να σας το πω και να το παλέψω, να πούμε τουλάχιστον ότι οι δαπάνες για ε, την παιδεία ε, ιδιωτική και δημόσια, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΩΣΑ, ε, θα πρέπει να φτάσουν στο 6%. Αυτές τις στατιστικές θα σας τις μοιράσω στη συνέχεια. Πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης το έχουν πετύχει αυτό το 6% στις δαπάνες για την παιδεία, ιδιωτική και δημόσια, επαναλαμβάνω. Και να έχουμε μια κοινή τροπολογία ή δυνατόν 6% γίνεται και παραπάνω για να πούμε ότι μάλιστα εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται συγκεκριμένο στους στόχους. Κατά τα άλλα, έχουμε τις κλασικές πολιτικές διαφορές, κλασικές πολιτικές τοποθετήσεις. Ορισμένοι θέλουν κάποια πολύ ουσιαστική και συγκεκριμένη ρύθμιση και αγωνίζεται γι' αυτό και στη στρατηγική της Λισαβόνας να υπάρχει σχεδόν εγγύηση για δραματική συρρήκνωση της φτώχειας, για δραματική συρρήκνωση ε, της ανεργίας των νέων με στόχους και κάποιοι άλλοι λένε να βάλουμε γενικές κατευθυντήριες γραμμές και για τη φτώχεια τώρα ας μην το θίγουμε και πάρα πολύ και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, ανταποκρίνονται αυτές οι τροπολογίες και οι απόψεις στο πολιτικό φάσμα που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και στα πολιτικά κόμματα. Θα δούμε αύριο στην ψηφοφορία τι θα γίνει. Ως εισηγητής στη συνάντηση με τους Σκιώδης είπα ότι με πολλές από τις τροπολογίες θα μπορούσα να συμφωνήσω αν δεν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες ή πάρα πολλές κρατιστικές τροπολογίες. Ε, με τους συντηρητικούς πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ ιδεολογικά με μερικές τροπολογίες, ναι, με άλλες όχι. Περιμένω να δω τι θα πείτε στη συζήτηση, θα μου εδώ προ το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν. Ο κύριο ε, Στόλογιαν που είναι ο σκιώδη εισηγητή για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Πολύ, καλή ήταν, πολύ καλές ήταν οι συζητήσεις μου με τον ε, εισηγητή, αλλά και εντός της πολιτικής μας ομάδας. Προσπάθησα τα σχόλια που άκουσα να τα συζητήσω ε, κατά τις επαφές μου με τον κύριο Μάρτιν. Δεν θέλαμε οι στόχοι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξηθούν μέσω των τροπολογιών για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την απασχόληση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 75% ο για την, στόχο για την απασχόληση και υπάρχει μια τροπολογία για αύξηση στο 80%. Και φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό Είπαμε τουλάχιστον 75% ότι θα έπρεπε να υποβάλουμε ως τροπολογία. Συμφωνούμε με τον συμβιβασμό αυτό. Και τον υποστηρίζουμε. Οπότε, ως γενική θέση προς τις τροπολογίες αυτές, είμαστε κατά της αύξησης ε, των στόχων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ακόμη ορισμένα σχόλια για, για παράδειγμα, σε μια τροπολογία αναφερόμαστε στην έννοια της οικολογικής ένωσης. Για μας είναι σαφέστατη η έννοια αυτή. Υπάρχουν και άλλες έννοιες που εμφανίζονται στα έγγραφα των ευρωπαϊκών οργάνων. Πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε ορολογία που είναι πλέον αποδεκτή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά και εκτός αυτών, για παράδειγμα, η Στρατηγική Ευρώπη 2020. Προτείνουμε αυτήν την έννοια της εφιούς ανάπτυξης, της περιεκτικής ανάπτυξης, και Πρόκειται για στόχου που πρότεινε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και τώρα λέμε μέσω μια τροπολογία ότι αντί για ευφυή ανάπτυξη θα έπρεπε να λέμε ευφυή διαχείριση της οικονομίας. Δεν συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι η διατύπωση Τη Στρατηγικής Ευρώπη 2020 που είναι περιεκτική, ευφυής και αϊφόρος ανάπτυξη είναι οι καλύτεροι όροι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στόλογεν. Στόλογιαν. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Λούντβικσον. Ευχαριστώ πολύ επειδή θα το ψηφίσουμε και έχουμε ήδη καθυστερήσει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Ήταν πολύ επικοδομητικός ε, ο εισηγητής. Ελπίζω, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε χρόνο, να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Ένα σχόλιο. Η εστίασή μας είναι η ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα αυτό θα μας βγάλει από την κρίση και μακροπρόθεσμα Έχουμε το στόχο της αηφόρου ανάπτυξης. Πρέπει όμως να έχουμε ποσοστά ανάπτυξης ε, λογικά που να λαμβάνουν υπόψη ε, το στόχο της αηφόρου, την αηφόρου ανάπτυξη. Όταν μιλάμε λοιπόν για την απασχόληση πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να υπάρξει ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο που ανέφερα. Δεν ε, έχει νόημα να είμαστε απλώς πολύ φιλόδοξοι στους στόχους μας. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ σε σχέση με το ποιου στόχου μπορούμε να επιτύχουμε. Αλλιώ θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη μείωση της φτώχειας ε, κατά 40% αντί για 25% όπως πρότεινε ο κύριος Μάρτιν. Θα έπρεπε να είμαστε ρεαλιστέ και ω προ το στόχο της απασχόλησης. 80% μου φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολικά φιλόδοξο. Ίσως ο συμβιβασμό που προτάθηκε προηγουμένω να είναι καλύτερο. Και οι γυναίκες και οι άντρε θα έπρεπε να έχουν την ίδια πρόσβαση, πρόσβαση στην απασχόληση. 62% είναι το ποσοστό για τις γυναίκες σήμερα και το να φτάσουμε το 80% μου φαίνεται λίγο... όχι ιδιαίτερα ρεαλιστικό. Θέλουμε όμως το στόχο και οι άνδρες και οι γυναίκες να έχουν ένα ε, ίσο επίπεδο απασχόλησης στο μέλλον. Άλλωστε αυτό είναι και ένα στόχος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτό, έχουμε πολύ περισσότερη δουλειά να κάνουμε σε σχέση με το ότι κάνουμε ε, σήμερα, δηλαδή να έχουν οι γυναίκες τις ίδιες ευκαιρίες στην αγορά απασχόλησης όπως και οι άντρες. Τρία στοιχεία θα ήθελα να υπογραμμίσω σε σχέση με τις δικές μου τροπολογίες. Πρώτον, νομίζω ότι είναι κεφαλαιόδου σημασίας οι διαθερωτικές αλλαγέ στα κράτη-μέλη να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάπτυξη να σημαίνει ψηλά ποσοστά απασχόλησης. Δηλαδή, με περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, ε, κατά την ανάπτυξη. Ο ρόλο των ε, κοινωνικών εταίρων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των πολιτών. Τα οι, οι πολιτικές απασχόλησης ε, στα κράτη-μέλη μπορεί να είναι επιτυχής αν οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν επαρκώς σε όλη τη διάρκεια του κύκλου από τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης μέχρι την εφαρμογή των ε, ε, σχετικών πολιτικών. Η κοινωνική συνοχή και αυτή συνδέεται με την απασχόληση και είναι κάτι που είναι θετικό και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Γιατί μεγαλύτερη απασχόληση σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μείωση της πτώχειας και κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ λογική προσέγγιση. Ελπίζουμε λοιπόν σε ένα καλό αποτέλεσμα μετά τους συμβιβασμούς που έγιναν ε, αύριο στη ψηφοφορία. Στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώδης ε, της είναι ο Τόμας Χέγκρε, δυστυχώς σήμερα κολλείται και με παρακάλεσε να πω δύο λόγια εγώ εξ του σήμερα. Επιτρέψτε μου ευθύ εξ αρχή μια προσωπική παρατήρηση. Αν μιλάω πολύ γρήγορα να μου κάνει κανένα νόημα διερμηνής. Εντάξει, προ το παρόν. Μια προσωπική παρατήρηση λοιπόν. Με τρομάζει λίγο η ιδέα που σε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα παρόντες τόσο λίγοι συνάδελφοι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, και ποιο είμαι εγώ να το κάνω. Θα ήθελα να το πω όμως, με εκπλήσει αυτό, με τρομάζει. Σε τόσα πολλά έγγραφα της Ένωσης μιλάμε για την απασχόληση, για τους πολίτες που εκπροσωπούμε, για τη δημιουργία απασχόλησης να βρίσκουν δουλειά που να τους εξασφαλίζει εισόδημα οι Ευρωπαίοι και να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους. Ε, και ζητώ συγγνώμη, αλλά με εκπλήσει η ισχνή παρουσία συναδέλφων την ώρα που συζητάμε αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Γενικότερα τώρα. Να πω μερικά πράγματα για ορισμένες εξελίξεις που αφορούν ε, την αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια και τη χαρακτηρίζουν από το 2001 μέχρι το 2006 περίπου αυξήθηκε η συνολική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από 58,2 σε 58,9. Είναι πολύ μικρή αυτή η αύξηση. Από το 1997 μέχρι το 2006 από 22 εκατομμύρια πήγαν σε 32 εκατομμύρια εκείνοι που δουλεύουμε σύμβαση ορισμένου χρόνου αυτό σημαίνει ότι γίνεται πιο επισφαλή η απασχόληση, δεν είναι μόνιμη η δουλειά. Η μερική απασχόληση πριν από 12 χρόνια ήταν 32 εκατομμύρια, τώρα είναι 40 εκατομμύρια στην Ευρώπη μερικώ απασχολούμενοι. 31 εκατομμύρια ε, αυτοαπασχολούμενοι, ανεξάρτητοι, πολύ συχνά είναι εκείνοι που δεν έχουν υπαλλήλου και είναι και πολύ ε, χαμηλόμιστοι. Και 17 εκατομμύρια περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία παρά από ε, το γεγονός ότι εργάζονται είναι φτωχοί. Δουλεύουν οι άνθρωποι, ε, είναι φτωχοί και δεν μπορούν να καλύπτουν τα μηνιαία τους έξοδα και ε, έχουν ανάγκη άλλα επιδόματα για να επιβιώσουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό, τι σημαίνει απασχόληση, τι σημαίνει κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, να μπορείς να ζεις από τη δουλειά σου. Πολύ μεγάλη ε, αυτή του Τόμας και της ομάδας μου και το τονίζω και θέλω να το πω ξανά γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα οι στρατηγικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγικές που πρότεινε και ακολουθούσε δεν βοήθησαν το να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Αυτή η επισφαλής μορφέ εργασία. το, λένε τα σκληρά στοιχεία σα τα είπα, αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα αυτά. Ο κόσμο δεν μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του, ακόμα και εκείνοι που εργάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο φιλόδοξοι στου στόχου μα για να αυξήσουμε την πολιτική πίεση, να γίνει κάτι στην απασχόληση, ε, οπωσδήποτε, ουσιαστικά. Καλή δουλειά καλές θέσεις απασχόλησης, ILO μιλάει για αξιοπρεπή δουλειά, decent work, ανθρώπινη δουλειά, να ε, συμμετέχει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά να βοηθάει και τον εργαζόμενο να επιβιώνει. Γι' αυτό θεωρώ επίσης σημαντικό και στην Οικονομική Επιτροπή να το θέσουμε αυτό, να το συζητήσουμε, αυτό το θέμα των φτωχών εργαζομένων, της επισφάλειας στην εργασία, της φτώχειας μέσα από την εργασία, δεν μπορεί να αφαιθεί μόνο στα χέρια της κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει και η οικονομική πολιτική να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μια τέτοια λοιπόν οικονομική πολιτική που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μπορεί ο κόσμος να δουλεύει και να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στρέζεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, ομάδας ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θα ήθελα να σας μεταφέρω τα σχόλιά μας για το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταλαβαίνουμε βεβαίω ότι κάθε μέλος της Επιτροπής αυτής ενδιαφέρεται να υπάρχουν όσο το δυνατόν ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Όμως είναι κατά τη διαφορετική η άποψή μα από αυτή που περιέχεται στι διάφορε τροπολογίε, γιατί πιστεύουμε ότι η απασχόληση, οι θέσει απασχόληση προέρχονται όχι από τι κυβερνήσει των κρατών μελών, αλλά από τι εταιρείε κυρίω, από τι επιχειρήσει. Και συνεπώ, η βασική μα θέση είναι ότι οι επιχειρήσει πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία. Πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη πίεση από που να προέρχεται από κανονισμούς και νομοθεσία. Συνήθως, η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και δεν έχει πάντοτε διασυνοριακή διάσταση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δίνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο στις επιχειρήσεις τους ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ελευθερία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος, ο πιο βέβαιος τρόπος για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Συμφωνούμε βέβαια με τους συναδέλφους ε, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τεράστιες επενδύσεις ε, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση των πολιτών τους, γιατί η κατάρτιση είναι ο σωστός τρόπος. Η ανάπτυξη όλο και περισσότερων ε, δεξιοτήτων. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες που ζητούν από τα κράτη-μέλη τη μεταρρύθμιση των κοινωνικών συστημάτων τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν φθηνότερα και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να δίνουν και κίνητρα στους ε, πολίτες να ε, βρίσκουν δουλειά, να εργάζονται και όχι να επαφίενται, να στα ε, επιδόματα, στα κοινωνικά επιδόματα. Εντελώς απαράδεκτη θεωρεί την ιδέα της οικολογικής απασχόλησης η δική μας ομάδα Πιστεύουμε ότι είναι ένας ευσεβής πόθος ε, εντελώς ε, εκτός πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Αν όχι, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρτιν να συνοψίσει τη συζήτηση. Uh, ναι. Μη μου θυμώσετε, αλλά επειδή είναι τόσο λίγοι παρόντες, θέλω να ρωτήσω κάτι, Το προλύσατε. Ποιο άρθρο αναφέρατε, αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο άρθρο, γιατί δεν το άκουσα. Σε ποιο παράγραφο αναφέρεστε συγκεκριμένα. να ε, το Ναι. Εκεί που γίνεται λόγος για την οικολογία και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Μάλλον χάθηκε ο αριθμός του άρθρου. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Όντως είναι μικρή η παρουσία των συναδέλφων. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να κάνω την εξής παρατήρηση, το προλαλήσατε. Ως εισηγητής, συμμερίζομαι σχεδόν όλες τις τροπολογίες σας. Είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ σαφής. Ε, σε μία όμως διαφωνώ και θα έλεγα να την καταψηφίσουμε. Ταυτόχρονα όμως βλέπω πάρα πολλές τροπολογίες από την πολιτική αριστερά που πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση με τις δικές σας. Υπάρχει ευρεία συνένεση και θέλω να τελειώσω απευθύνοντας μια έκκληση. Βέβαια οι πράσινοι απουσιάζουν. Τι γίνεται με τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, αν θέλουμε ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, πώς μπαίνει εκεί η οικολογία. Εκεί συμφωνώ με την αριστερά, αλλά αν έχουμε λιγότερες ιδεολογικές παροπίδες και δούμε πιο υφάλαια, τι δυνατότητες έχουν με την κρίση τα κράτη, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε και γέφυρες μεταξύ ε, συντηρητικών εντό εισαγωγικών και αριστερών ε, διεξόδων. Στο βαθμό που δεν είναι τα πάντα νέο φιλελεύθερα ή τα πάντα απέτηση να τα χορηγεί το κράτος. Ελπίζω τελικά να βρεθεί πολιοψηφία και να υπερψηφιστεί η έκθεση. Με ευχαριστώ. Um, Μάλιστα. Η ψηφοφορία είναι αύριο στις 22 Ιουνίου και στην αρμόδια επιτροπή 14 Ιουλίου. Και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, κατά πάσα πιθανότητα, την 1η Σεπτεμβρίου. draft opinion. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Νομικών προσωρινά μέτρα σχετικά με το πάχωμα και τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του φιλέτη στι διασυνοριακές περιπτώσεις. Ο κύριος Τόλος αν έχει το λόγο, εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών ε, Θεμάτων την οποία χαιρετίζουμε. Γιατί στην ενιαία αγορά όταν γίνεται όταν γίνονται οικονομικές συναλλαγές δεν λαμβάνουν πάντοτε την αμοιβή τους βάση των συμβάσεων που έχουν υπογράψει. Και επειδή όλο και περισσότερες διασυνοριακές ε, ε περιπτώσεις ε, εμφανίζονται, πιστεύουμε ότι έτσι θα ενισχύσουμε την ε, ακεραιότητα και την συνέπεια της ενιαίας αγοράς και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε νομοθετικά μέτρα με σκοπό να εναρμονίσουμε τις πηγές πληροφοριών από τα κράτη-μέλη που είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να είναι διαφανή, διαθέσιμα, προσβάσιμα και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν ένα συμβαλόμενο μέρος δεν ε, πληρεί τι ε, συμβατικές του υποχρεώσεις, ε, τότε το συμβαλόμενο αυτό μέρος, όταν δεν δίδει πληροφορίες για τα περιουσιακά του στοιχεία, πριν να φτάσουμε στο δικαστήριο, είναι καλύτερο να αναπτυχθούν τα μέτρα τα οποία προτείνουμε. Τα μέτρα επίλυσης των διαφορών που προέρχονται από εμπορικές συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται προσπάθειες ε, επίλυσης διαφορών μεταξύ του οφηλέτη και του αντισυμβαλωμένου μέρους και σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν σε κάποια συνεννόηση τα συμβαλώμενα μέρη για την αποζημίωση. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας τέτοιο είδους μηχανισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τυποποιήσουμε δηλαδή τους ε, τρόπους με τους οποίους ε, μπορεί να ε, επιλύεται η διαφορά μεταξύ των μερών και των οργανισμών επιβολής της νομοθεσίας σε περίπτωση συμβάσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια τυποποίηση. Το ίδιο είχαμε κάνει και κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, τυποποίηση των τρόπων ανάκτησης χρέους στους ε, οργανισμούς ε, των κρατών μελών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Για να ενισχύσουμε ακριβώς τη συνεργασία των μηχανισμών επιβολής ε, στα κράτη-μέλη που ε, είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά και με τις ένομες τάξεις προκειμένου να επισπεύσουμε την ανάκτηση του χρέους Και πιστεύουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε και εκείνη σύντομα να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία σε σχέση με το θέμα αυτό πριν από το 2013. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στόλογιαν. Ο κύριος Κλούτε από τους σκιώδεις εισηγητές. Να αρχίσουμε με εσάς κύριε Κλούτε. Ναι, ευχαριστώ. Τώρα βέβαια εγώ δεν έχω προετοιμαστεί γιατί δεν είμαι ισχυώδης ηγητής και δεν θέλω να σας φάω το χρόνο, παρετούμε, δεν έχω να πω τίποτα. Okay, uh, Καλώς. Η Αρλίν Μακάρθε είναι σκιώδης συγγήτρια, αλλά και συγγήτρια στην Επιτροπή, επί της ουσίας στην Νομική Επιτροπή και μου ζήτησε να διαβάσω το εξής εξ ονόματός της. Καθορίζει τη δυνατότητα εκπόνησης θέσης του Κοινοβουλίου σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εκατομμύρια επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το δικαίωμα ε, εμπορικών συναλλαγών στην εσωτερική αγορά εκατομμύρια πολιτών ε, χρησιμοποιούν το δικαίωμα να ζουν και να ταξιδεύουν ε, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βασικό στοιχείο της εργασίας μας να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν ε, δικαιώματα για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Σε περίπτωση τέτοιων διασυνοριακών χρηματικών απαιτήσεων θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα επιβολής αμοιβαία αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων όπως είναι το αντίστοιχο διάταγμα ε, για τις διαδικασίες πληρωμών, για τις διάφορες αξιώσεις κτλ. Ωστόσο, ε, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στη διαδικασία ε, με την απόφαση και μόνο, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά. Αυτό προ όφελο των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα βασικό στοιχείο τη αποτελεσματική επιβολή και υιοθέτηση των αποφάσεων είναι τα δικαστήρια να μπορούν γρήγορα να ζητούν πρόσβαση ε, στις, ε, στα στοιχεία, την περιουσία και πάγωμα των στοιχείων. Ε, αλλιώς κάποιοι κακόβουλοι και παρανομούντες μπορούν να μεταφέρουν τα περιουσιακά του στοιχεία αλλού σε άλλη δικαιοδοσία και να είναι ένα βήμα μπροστά από τον νόμο. Και ο πολίτης που ε, ψάχνει το δίκιο του θα δαπανίσει πολύ χρόνο και πολλά χρήματα και μπορεί να χρειαστεί να πάει και σε άλλο κράτος μέλος, σε άλλα δικαστήρια για να δικαιωθεί χωρίς καμία εγγύηση ότι θα ανακτήσει το χρέος, ότι θα έχει κάποια ε, επιτυχή έκβαση. Γι' αυτό χρειάζεται ε, σαφής ε, ρύθμιση ε, για το άνοιγμα των λογαριασμών, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτές που να ζητούν το λόγο επ' αυτού, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα κύριε Στόλογιαν ε, συμπερασματικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η γραμματεία της Επιτροπής, η Επιτροπή τέλος πάντων, ζήτησε μια παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των τροπολογιών. Ε, νομίζω ότι το Σεπτέμβρη έχουμε, είχαμε βάλει μια προθεσμία. Επομένως θεωρώ ότι έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στο σχέδιο αυτό της έκθεσης. Και εδώ απευθύνομαι σε όλες τις ομάδες, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει χώρος βελτίωσης. Ευχαριστώ κύριε Σαλαζάν. Όντως 12 της 7 η Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Επομένως έχετε δίκιο, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας ενημερώσουμε με email για την συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η συζήτηση των τροπολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή έχει σχεδιαστεί, έχει προγραμματιστεί για τις 5 ε, Οκτωβρίου, ενώ στην άλλη Επιτροπή θα έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία τέλος Νοεμβρίου. στην Επιτροπή για τα νομικά θέματα. Τώρα, επειδή στις 4.30 θα έρθει ο κύριος Τρισέ, θα διακόψουμε την συνεδρίαση για λίγα λεπτά, 11 λεπτά συγκεκριμένα, και μετά θα ξαναρχίσουμε. Μήπως θα μπορούσατε να καθίσετε για να συνεχίσουμε. And then eventually we will let the photographers go. Θα μπορούσαν να αποχωρήσουν οι φωτογράφοι. Hey. Okay. Uh take Να το επαναλάβω, να καθίσετε για να συνεχίσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι καλωσορίζω τον κύριο Τρισέ για τον τακτικό μας διάλογο για τα δημοσιονομικά. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η συνήθις. 15 λεπτά θα μας μιλήσει ο κύριος Τρίσε και μετά ο καθένας θα έχει 1,5 λεπτό στη διάθεσή του για να κάνει ερώτηση και 3 λεπτά ο πρόεδρος για να απαντήσει. Επομένως γίνεται επίσης και μια κατανομή του, του χρόνου ομιλίας ε, ανάλογα με τις ομάδες. Ξέρετε τον, ε, τον τρόπο και την ε, μέθοδο που θα ακολουθήσουμε. Ε, το λόγο θα τον πάρουν όλοι οι συνάδελφοι ανάλογα με την δύναμη της ομάδας τους. Δεν είναι μια διαδικασία κάτσο διάη. Λοιπόν, ε, καλωσορίζω για άλλη μια φορά τον κύριο Τρισέ και ελπίζω ότι οι φωτογράφοι μόλις ξεκινήσει να μιλάει θα αποχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη από την τελευταία μας συνάντηση 22 Μαρτίου, η Ευρωζώνη αντιμετώπισε μία από τις πιο προκλητικές περιόδους της από την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις ε, χωρίς προηγούμενο ε, στις ε, οικονομικές αγορές. Οι δημόσιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υιοθέτησαν πολύ αυστηρά μέτρα. Πρόσφατα ελήφθησαν πολύ σημαντικές αποφάσεις και απαιτούν εξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που οπωσδήποτε ανακύπτουν και εδώ στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό καλωσορίζω τη δυνατότητα που μου δίνεται να έχουμε αυτή την ανταλλαγή και με τη σημερινή ακρόαση όλος ιδιαίτερους χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία. Να ξεκινήσω την παρέμβασή μου ως συνήθως κάνοντας μία αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης. Θα επανέλθω μετά στην απόφαση που εξεγγέλθη την, την 10η Μαΐου ε, να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις ε, στην αγορά των ομολόγων στην ζώνη του ευρώ και σε ένα τρίτο λόγο θα ασχοληθώ με τους μηχανισμούς οικονομικού συντονισμού της ε, ευρωζώνης και των, αλλαγό, των αλλαγών συγγνώμη, ε, που απαιτεί η παρούσα κατάσταση. Από την προηγούμενη ακρόση το Μάρτιο, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της ε, Ευρωζώνης ε, το πρώτο ήμιση του 2010. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ε, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% ανά τρίμηνο τους τρεις πρώτους μήνες του έτους αυτού και φαντάζομαστε ότι σύμφωνα με τις ε, προσδοκίες μας η οικονομία στην, ε, στην Ευρωζώνη θα διευρυνθεί ε, με τριοπαθώς αυτή τη χρονιά και οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται. Οι τελευταίες μας προβολές για το... στο ευρωσύστημα ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με αυτή την αξιολόγηση. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού για την Ευρωζώνη ήταν 1,6% τον Μάιο, αυξήθηκε κατάτι από το 1,5% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της υψηλής ε, τιμής ε, των, των, τιμών σε ενεργειακό τομέα. Επίσης, ε, Υπάρχει μια μικρή αύξηση στον πληθω... περιμένουμε μια μικρή αύξηση του πληθωρισμού στο δεύτερο ημίση του 2010. Οι νομισματικές μας αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις ε, μέσω πρόθεσμα θα παραμείνουν. Αυτό αντικατοπτρίζεται κυρίως ε, στην, ε, λόγω του ε, του της συνολικής ε, μικρής αύξησης ε, του χρήματος και των πιστώσεων. Ο, υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο πληθωρισμός δεν θα είναι οι, οι, οι διάφορες ε, παρατηρήσεις που γίνονται για τον πληθωρισμό και για ε, την εξέλιξή του θεωρούνται, θεωρούνται μάλλον αβάσιμε. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τον, ε, για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη φαίνεται ότι είναι θετικές, τουλάχιστον σύμφωνα με, με τον ορισμό της, που έχουμε για την σταθερότητα των τιμών. Λαμβάνοντα υπόψη τώρα τις, το τι προβλέπουμε όσον αφορά την σταθερότητα των τιμών και τις προσδοκίες για τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η νομισματική μας πολιτική και το παρόν επίπεδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το πλέον κατάλληλο. Τώρα, θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με την απόφαση του Δικητικού Συμβουλίου να παρέμβουμε στην ζώνη του ευρώ, για την, κυρίως όσον αφορά τα ομόλογα τις αγορές των ομολόγων. Κάτι το οποίο είχαμε ανακοινώσει στις 10 Μαΐου μετά την απότομη και την πολύ σημαντική μείωση στις εντάσεις των δημοσιονομικών αγορών σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως και στην Ευρώπη. Αυτές οι εντάσεις διευρύνθηκαν σε μεγάλα κομμάτια των χρηματοπιστωτικών αγορών, ακόμα και στην αγορά των μετοχών, στην διατραπεζική αγορά και στην αγορά ξένων, ε, ξένου συναλλάγματος. Είδαμε ποια ήταν η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε ε, τον Οκτώβριο του 2008 μετά την κατάρρευση του, της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, είδαμε ότι υπάρχει μια, ένα ευμετάβλητο στις αγορές, ευμετάβλητο το οποίο ε, εντάθηκε ε, όχι μονάχα όσον αφορά τις αγορές των κρατικών ομολόγων, αλλά και στις χρηματαγορές. Ε, οι συναλλαγές ε, στην διατραπεζική αγορά μειώθηκαν σημαντικά και επικρατεί μια βεβαιότητα ανάμεσα στις τράπεζες όσον αφορά την φερεγγιότητα των ομολόγων τους. Ε, αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα των τραπεζών που είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη για να προσφέρουν επίστοση στην πραγματική οικονομία μπορεί να πληγεί σημαντικά. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξήγηλε στις 10 Μαΐου όχι μόνο την επανεργοποίηση, την επανεργοποίηση του, των ε, προηγούμενων μέτρων, αλλά επίσης και την επανεργοποίηση των συμφωνιών SWAP με, την, ε, με το Federal Reserve, αλλά επίσης και την παρέμβασή της στις αγορές των ομολόγων με την ε, ενεργοποίηση του προγράμματος για τις αγορές των ομολόγων. Λοιπόν, η αγορά, οι κρατικές αυτές αγορές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τρεις λόγους. Καταρχάς, τα επιτόκια ε, των κρατικών ομολόγων θέτουν ένα όριο για τα επιτόκια τα οποία οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν όταν εκδίδουν τα ομόλογά τους. Ε, εφόσον οι αγορές είναι διαταραγμένες, τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορούν να, δεν μπορούν να μετακυληθούν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και επομένως οι τιμές και στις τιμές ε, αυτό είναι που, αυτό το οποίο ονομάζουμε κανάλι τιμών, the price channel. Κατά δεύτερο λόγο, εάν έχουμε χαμηλότερες τιμές ομολόγων, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλότερα επιτόκια που συνδέονται με τις διαταραγμένες αυτές αγορές ομολόγων, το οποίο κάτι το οποίο θα δημιουργήσει σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια του χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Για τις τράπεζες αυτό θα περιορίσει την ικανότητά τους να προσφέρουν δάνεια στην οικονομία. Και τρίτον, ε, εάν έχουμε χαμηλή ρευστότητα για τα κρατικά ομόλογα ε, αυτό θα περιορίσει τον ρόλο τους σαν εγγύηση σε ε, συναλλαγές επαναχρηματοδότησης. Επομένως αποφασίσαμε να παρέμβουμε. Ο στόχος του προγράμματος δεν είναι να εγχύσουμε συμπληρωματική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Θέλουμε να εξουδετερώσουμε τις αγορές ομολόγων μέσω συγκεκριμένων συναλλαγών επαναρρώσεων ε, σαν αποτέλεσμα το επίπεδο ρευστότητας και τα επιτόκια στην αγορά, στις χρηματαγορές δεν επηρεάζονται από το πρόγραμμα αυτό. Με άλλα λόγια δηλαδή η νομισματική μας πολιτική δεν επηρεάζεται και δεν υπάρχουν κίνδυνοι πληθωριστικοί που να συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα να τονίσω ότι πήραμε αυτή την απόφαση να εισάγουμε το πρόγραμμα αυτό για τις αγορές των ομολόγων ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με τις, συνθήκες, με τις ε, διατάξεις της συνθήκη Επίσης, ε, ε, επίσης ε, υιοθετήσαμε τις δεσμεύσεις αυτές με απόλυτη ανεξαρτησία. Συνειδητοποιούμε ποιε είναι οι δεσμεύσει ε, που υιοθέτησαν ε, οι κυβερνήσεις ε, της Ευρωζώνης πριν από, το, από εκείνο το Σαββατοκύριακο, την, την παραμονές της Παρασκευής 7 Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την δήλωση που έκαναν οι κυβερνήσει της Ευρωζώνη ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ικανοποιήσουν του στόχου, του στόχους αυτής της χρονιάς και των επομένων ετών, ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις διαδικασίες για το υπερβολικά ελλείμματα και ε, θα υιοθετήσουν ε, ε, συμπληρωματικές δεσμεύσεις κάποιες τουλάχιστον κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έτσι ώστε να επιταχυνθεί η φορολογική ενοποίηση και να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Εδώ θα περάσω στο τρίτο θέμα μου γιατί μου ζητήσατε κυρία Πρόεδρε να μιλήσω για, την ενισχυμένη, τον ενισχυμένο οικονομικό συντονισμό και επίβλεψη στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι η ότι χρειάζεται να γίνει ένα άλμα μέσα στα πλαίσια της επίβλεψης και της προσαρμογής των φορολογικών ε, πολιτικών. η de facto αλληλεγγύη την οποία, την οποία ζήτησε ο Ρομπέρ Σουμάν πριν από 60 χρόνια αντικατοπτρίζεται σε ένα βαθμό στην οικονομική ε, ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση που, την, οποία έχουν, την οποία έχει πετύχει η Νομισματική Ένωση. Αλλά η αλληλεγγύη είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Τα πλεονεκτήματα και η προστασία που προέρχονται από τη συμμετοχή στην Νομισματική Ένωση επιβάλλουν επίσης και υποχρεώσεις και ευθύνες. Επομένως τώρα θα πρέπει να έχουμε με μια πιο ε, αποτελεσματική δομή για φορολογική μακροοικονομική επίβλεψη και προσαρμογή. Με βάση τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Task Force υπό την προεδρία της, ε, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Βαν Ρόμπ Ρόμπεϊ, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο βασικούς ε, τομείς μεταρρυθμίσεων. Ένας τρίτος τομέας ε, που είναι το πλαίσιο ε, διαχείρισης των κρίσεων εξετάζεται ακόμα σε επίπεδο task force. Λοιπόν, καταρχάς, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η επίβλεψη των φορολογικών πολιτικών πρέπει να ενισχυθεί ε, και μπορώ να σας πω με μεγάλη μου χαρά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε αυτή την ε, αξιολόγηση στην συνάντηση που είχε την προηγούμενη Πέμπτη. Στο επίπεδο των 27 και πιο συγκεκριμένα και στην, στο ιστορικό της Ευρωζώνης έχουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να προλάβουμε και να διορθώσουμε ή δυνατόν και εφόσον είναι απαραίτητο τα υπερβολικά ελλείμματα και τα επίπεδα του χρέους. Μια πιο αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών είναι απαραίτητη. Επίσης, η φορολογική δημοσιονομική επίβλεψη πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και άμεση. Πρέπει να στηρίζεται σε πιο ανεξάρτητη το έλεγχο και αξιολόγηση. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση όσον αφορά την επίβλεψη ανάλογα με τις ε, επιδόσεις κάθε κράτους, κάθε κράτους. Η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευθύνη στην υποβολή προτάσεων που μπορούν να τροποποιηθούν με ομοφωνία στο Συμβούλιο και να μην κάνει μόνο συστάσεις με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις πολύ νωρίτερα και να είναι πολύ ευρύτερες. Ε, δεν θα πρέπει να αφορούν οι κυρώσει αυτές μόνο το, υπερ, ε, το υπερβολικό χρέος και την αναλογία υπερβολικού χρέους, αλλά να επιβάλλονται και όταν οι χώρε δεν κάνουν επαρκή, δεν, ε, επαρκή βήματα για να πετύχουν μια διόρθωση, αν θέλετε, των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών του στόχων ένα ευρύτερο φάσμα ε, κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με μη, οικονομικά, ε, με, πιο, οικονομικές και διαδικαστικές κυρώσεις. Αυτό ο δεύτερο τομέα μπορεί να φαίνεται πιο καινοτόμο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τονίσει το θέμα αυτό στο Eurogroup από το το, από το 2005 τουλάχιστον η επίβλεψη των πολιτικών, ε, η παρακολούθηση των πολιτικών για να διατηρηθεί η εσωτερική και εξωτερική ανταγωνιστικά της Ευρώπης, οι πολιτικές για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, για να ενισχυθούν τα, τα ικανότητες των ανθρώπων και για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι τομεί που μας αφορούν. Αυτές οι πολιτικές ξεπερνούν, αν θέλετε, το, τον τομέα του, του εμπορίου. Συμπεριλαμβάνουν ναι, και τους υπόλοιπους τομείς, τον δημόσιο τομέα κυρίως, μια και είναι τόσο αποφασιστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο σύνολό της ένα, μια συνειδητή διαχείριση των μισθών και του, και του, και του κόστους έτσι ώστε να, διατηρηθεί μια υγιής θέση ε, για την οικονομία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος για μια πιο ευρύτερη μακροοικονομική επίβλεψη. Ο λόγος για τον οποίο η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος μας ε, δεν είναι επειδή οι χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν μια πολιτική που να στηρίζεται και να προσανατολίζεται στην, στις εξαγωγές ή για να ενισχύσουν το, διεθνές τους, το μερίδιο στη διεθνή αγορά. Ο λόγος είναι ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχετική ανταγωνιστικότητα των οικονομιών στηρίζεται κυρίως και, και στηρίζει με τη σειρά του την βιωσιμότητα των τιμών και, του κόστους. Χαίρομαι διότι την ε, προηγούμενη Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επίβλεψης στον τομέα αυτό. Η εμπειρία μας έδειξε ότι, ότι αν υπάρχουν ε, ε, διαφορές συνεχείς μεταφορές, διαφορές γνώμη, αυτό σε αυτό τον τομέα. Αυτό είναι εις βάρος και των κρατών μελών και της Νομισματικής Ένωσης στο σύνολό της. Θα πρέπει επομένως να επιτρέψουμε να γίνονται επίσης και στοχευμένες και διαφοροποιημένες ε, παρακολουθήσεις ή επιβλέψεις και να υιοθετούνται μέτρα παρακολούθησης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στηρίζονται ε, στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων και από την Κομισιόν και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι εμπειρογνώμονες αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή ε, τρόπους για να λάβουν υπόψη τον περίπλοκο του τομέα αυτού και εάν μπορούμε να υιοθετήσουμε αποτελεσματική, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επίβλεψης και προσαρμογής και όσον αφορά τις ε, δημοσιονομικές και όσον αφορά τις, ε, ανταγωνι... Ε, πολιτικές ανταγωνισμού και αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσω μιας σωστής νομοθεσίας το, το γεγονός ότι το δημοσιονομικό μας σύστημα εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία και όχι το ανάποδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα, θα ξεπεράσουν την κρίση αυτή και θα γίνουν δυνατότερες θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι μια και χανάζουμε μια πορεία ανάμεσα αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να εργαστούμε όλοι σκληρά και να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις ανάλογα με την, που να είναι ανάλογες με την σημασία της Ένωσης. Εμείς είμαστε μια ενιαία αγορά 500 εκατομμυρίων πολιτών και έχουμε μια οικονομική και νομισματική ένωση 330 εκατομμυρίων πολιτών. Επομένως, οι, αυτοί οι οποίοι χαράζουν την πολιτική πρέπει να λάβουν υπόψη ακριβώς την ε, ε, ανάγκη να εξυπηρετήσουν τους πολίτες αυτούς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ε, φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Η αντίδραση της Ευρώπης σε χρόνους κρίσης είναι να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνοχή. Και θα ήθελα να σας ζητήσω, σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σαν εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης, να συνεχίζετε να μας στηρίζετε στο δρόμο που έχουμε χαράξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρίσε. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις, σε ερωταποκρίσεις. Την περασμένη φορά είχαμε αποφασίσει ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε την ερώτηση και την απάντηση. Αλλά θα έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας, μερικά λεπτά για την απάντηση. Και επίσης ε, θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής να μην, ε, κάνουν τεράστιες παρεμβάσεις. Πρώτα, ο Ζων Πολ Κοζές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτήν την δύσκολη περίοδο κρίσεως. Μιλήσατε για πολλά ζητήματα. Το συμπέρασμά σας ήταν ότι μπορείτε να υπολογίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Όντως, ε, δεν ε, δεν ε, υπάρχουν οι υπέρ, οι υπέρ και οι κατά. Δεν θα σας πω που βρίσκονται οι κατά, αλλά οι υπέρ βρίσκονται σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν βέβαια χώρε ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Αναφερθήκατε και εσεί στο είδο των υποχρεώσεων των ε, ε, Ευρωπαϊκό, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που, που δεν είχε στο παρελθόν αλλά έχει τώρα. Μιλήσατε για τι πληθωριστικές πιέσει, μήπως θα μπορούσατε να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένο προ αυτό και ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την έξοδο από την κρίση και τι θα γίνει μετά την έξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Όσον αφορά το ερώτημα για τον πληθωρισμό, όπως ανέφερα και στην ε, ομιλία μου, ευρώ προς ευρώ ανακτούμε την, ε, ε, την ρευστότητα που έχουμε στο πλαίσιο του προγράμματός μας και το είπαμε και στην, στις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούμε ότι είναι ότι η νομισματική πολιτική είναι η σωστή, πιστεύουμε ότι τα επιτόκια είναι τα κατάλληλα και δεν αλλάξαμε την νομισματική μας ε, πολιτική. Συνεπώς ε, εξουδετερώσαμε το νέο αυτό μη συμβατικό ε, πρόγραμμα και ε, όπως είπα καταφέραμε να ανακτήσουμε ό,τι δώσαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. 47 δισεκατομμύρια ευρώ είχαμε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα φέτος, ε, αυτή την εβδομάδα 47 συν 4. Τα επιπλέον 4 ε, είναι για να αντισταθμίσουν ε, αυτά που είχαμε κάνει την προηγούμενη, την ε, αντιπροηγούμενη εβδομάδα. 47 συν 4, 51. Και θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε αυτά τα ποσά ευρώ προς ευρώ. Όπως και κάθε πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν συμβατικό και είχε αποφασιστεί, Βεβαίω έχει μία περιορισμένη διάρκεια, αλλά δεν ε, θα ήθελα να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή και δεν θα πω και περισσότερα όσον αφορά τις ε, αγορές ε, για τις οποίες παρεμβαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εδώ κάθε φορά που πάνε άσχημα τα πράγματα, ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να ε, τονώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι λένε ότι χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση. Τι είναι αυτή η οικονομική διακυβέρνηση, κανείς δεν γνωρίζει. Ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για το άρθρο 121-136, ο πρόεδρος Σαρκοζή για μια κυβέρνηση της Ευρωζώνης αρχή κρατών και κυβερνήσεων. Η κυρία Μέρκελ καγκελάριο λέει όχι της Ευρωζώνης αλλά της Ένωσης Οικονομική Κυβέρνηση. Λένε ότι προηγουμένως θα πρέπει να χαλιναγωγηθούν οι υπολογισμοί και να σεβόμαστε τις εθνικές διαδικασίες. Η καγκελάριο Μέρκελ λέει θα πρέπει να αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου από εκείνους που δεν συμμορφώνονται. Η Ισπανική Προεδρία λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Εσείς λέτε να επιβληθούν κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές πρόθεσμα. Δίνουμε λεφτά στην Ελλάδα, θα τις θα πάρουμε με το άλλο χέρι ως κυρώσεις οικονομικές. Όταν μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα, συμφωνούμε ότι η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού ε, δεν έχει δώσει αποτελέσματα. Χάσαμε ανταγωνιστικότητα σε καλούς καιρούς βγαίνουμε πιο αργά από την κρίση από ό,τι κάποιοι άλλοι, χρειάζεται διόρθωση αυτό. Πώς θα αλλάξουν αυτά, πώς θα τροποποιηθούν και πώς θα περάσουμε τώρα από τη φιλολογία στην πράξη. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να δεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι το γράμμα και το πνεύμα του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας δεν έχουν γίνει πλήρως σεβαστά. Αυτό το λέω επανελειμμένα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωρίζω ότι συμφωνεί και το Κοινοβούλιο. Αυτό μας λυπεί όλους. Ήταν πολύ λυπηρό και νηλημένα έχω πει ενώπιόν σας ότι μπορεί να έχουμε ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν έχουμε πλήρη ομοσπονδιοποίηση. Χρειαζόμαστε το αντίστοιχο ενός ισχυρού πλαισίου το οποίο δεν διαθέτουμε γιατί δεν έχουμε πολιτική ομοσπονδία με ε, τα όργανα και τους θεσμούς της. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πάλι μας έχει δείξει εμπειρία ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. Τώρα το γνωρίζουμε ακριβώς επειδή έχει αυτή την ένταση που έχει η κρίση ότι δεν θα έπρεπε μόνο να γίνει πλήρω σεβαστό το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη. και γνωρίζετε ότι τότε κάποιες χώρες προσπάθησαν να αποφύγουν το πλήρη σεβασμό του Συμφώνου και τη σωστή εφαρμογή του. Όχι μόνο λοιπόν αυτό, αλλά και μετά από την εμπειρία που έχουμε πλέον με τη σημαντικότερη κρίση που έχουμε ζήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μιλώ και για κρίση στη λειτουργία μας, θα πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο αυτό. Πολύ περισσότερο, κατά την άποψή μας, από εκείνο που ήταν το σύμφωνο σταθερότητας και Ανάπτυξη στην αρχή. Μιλούμε για ένα ε, ποιοτικό άλμα, κφαντικό ποιοτικό άλμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, απαντώ, έχω και προβλήματα χρόνου. Ως εξή την ερώτησή σας. Ως ένα πρώτο βήμα Η δευτερογενής νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται πλέον, και μάλλον να εφαρμόζουμε ό,τι μας επιτρέπει η δευτερογενής ε, νομοθεσία πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και τι είναι εδώ. Πρόληψη, ε, νομισματική εποπτεία, κυρώσεις, αυτοματισμό κυρώσεων που είναι επιθυμητό, Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι μας επιτρέπει η νομοθεσία θέλουμε να το κάνουμε. Και σε ένα δεύτερο χρόνο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μήπως χρειάζεται τροποποίηση τη συνθήκη. Αλλά σαν ένα πρώτο βήμα, ό,τι μας επιτρέπει δευτερογενή νομοθεσία χωρίς αναθεώρηση τη συνθήκη, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την άποψή μα. So everything. Uh, δηλαδή, η κυρία Κράτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σε παλαιότερη συμμετοχή σας σε συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τον περασμένο Μάρτιο, μας είχατε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίζει να αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα ε, χωρίς ε, ε, προϋποθέσεις της βαθμολόγησης και αξιολόγησής τους. Οι τελευταίες όμως εξελίξεις μας βάζουν σε προβληματισμό. Είχαμε την υποβάθμιση από τη Moody's, ε, με τις ε, αντιδράσεις των Ευρωπαίων εξωματούχων χαρακτηρίζοντάς τη σαν μια ατυχή απόφαση κυρίως στην κρίσιμη συγκυρία που βρίσκεται η Ελλάδα και από την άλλη μεριά δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα επιβάλλει την πρόσθετη χρέωση το haircut το 5% στα ελληνικά ομόλογα. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς αυτό αν αληθεύει, δεύτερον πώς εκτιμάτε ε, την ε, επίπτωση ενός τέτοιου μέτρου στην ε, ανάγκη, στην κρίσιμη ανάγκη ρευστότητας που έχει η Ελλάδα και τις συνέπειες που θα είχε σε ρευστότητα αυτό το μέτρο και δεύτερον πόσο οι αξιολογήσει των διεθνών οίκων επηρεάζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Όπως ξέρετε, είπαμε εκ των προτέρων για τα κρατικά ομόλογα ότι θα εξετάσουμε την ε, επιλεξιμότητά τους όσον αφορά το, την εγγύηση, αν θέλετε, τα χέγγια, ανεξάρτητα, ανεξάρτητα από την βαθμολογία τους. Και αυτό είναι τα κρατικά. Μιλάω μόνο για τα κρατικά ομόλογα. Και επιτρέψτε μου να σας πω τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα τελευταίο, τελευταίο καιρό τέλος πάντων, κυρίως το πρόγραμμα ανάκαμψης ε, το οποίο εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις ε, ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις ε, που πήραμε και στην Αθήνα και για το πρόγραμμα προσαρμογών αλλά και στο το Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και τις αποφάσεις που ληφθήσαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η κατάσταση σήμερα αντικειμενικά είναι καλύτερη όσον αφορά την σοβαρότητα και την σταθερότητα του ελληνικού προγράμματος σε σχέση με τον καιρό που δεν είχαμε ούτε πρόγραμμα και ούτε αποφάσεις ελληνικής κυβέρνησης ε, να προχωρήσει στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ε, και δεν είχαμε αποφάσεις ούτε στη Ουάσιγκτον ούτε στις διάφορες ευρωπαϊκές ε, πρωτεύουσες. Και ούτως ή άλλως τότε η βαθμολογία ήταν καλύτερη όταν αντικειμενικά η οικονομία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι τώρα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Σταματώ εδώ, δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Thank you. Uh, Edward Ευχαριστώ, Edward Cicluna. Uh, Κύριε Τρισέ, θυμάμαι ότι είπατε ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα η Ευρωζώνη, αλλά τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν όντω ισχύει αυτό, δεν νομίζετε ότι χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα των τεστ κοπόσεων των τραπεζών που υπάρχουν, τα ακούσαμε και στα νέα, αλλά και την ανταπόκριση των κρατών μελών ανάλογα με τα διάφορα σενάρια που μπορεί να ισχύσουν. Και Πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν εγγενή προβλήματα ε, στην Ευρωζώνη ε, ως προς το ε, κοινό νόμισμα και πιστεύετε ότι ό,τι έχουμε κάνει είναι επαρκές για να προλάβουμε τις μελλοντικές κρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αν είχε εφαρμοστεί αυστηρά το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα ήμασταν σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτού. Τώρα, το κατά πόσο θα ήμασταν σε μία κατάσταση δεδομένης βέβαια της ε, ε, έντασης της κρίσης ε, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, κατά πόσο λοιπόν θα βρισκόμασταν σε μια ε, κατάσταση στην οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε περιβάλλον πλήρου σταθερότητα, πολύ αμφιβάλλω. Πρέπει και εμεί ε, να μάθουμε το μάθημά μα από την κακή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα και ε, Ανάπτυξη, αλλά επίση να δούμε και τι είναι πραγματικά αυτό το τεστ κοπόσεω το οποίο πρέπει να κάνουμε, ε, πρέπει να περάσουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ένα ποσοτικό άλμα για την, προς την εποπτεία Πιστεύω ότι θα το μετανιώσουμε πάρα πολύ αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να κινηθούμε προς την επιτήρηση, την εποπτεία ε, των ε, δημοσιονομικών πολιτικών αλλά και των δικτών ανταγωνιστικότητας ε, που πάντοτε εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο ενιαίου νομίσματος. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει και να βελτιώσουμε την εποπτεία αλλά και το συντονισμό σε επίπεδο των 27 κρατών μελών. Νομίζω ότι υπάρχει και το επίπεδο των 27 κρατών μελών. Είμαστε μια ενιαία αγορά. Μια ενιαία αγορά είναι μια οντότητα που είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί σωστά και βεβαίως εντός ε, των 27 πρέπει να ενισχύσουμε την εποπτεία των 16 που μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σάντσε Πεσέντο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρισέ, θα ήθελα να σα συγχαρώ. Να σας συγχαρώ, λέγω, για το έργο σας τους τελευταίους μήνες. Πολύ θετικό νομίζω ήταν για την Ένωση. Σε σχέση με τη δημοσιονομική υποπτία και την ανταγωνιστικότητα στην οποία αναφερθήκατε, υπάρχει το εξή πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να συνδεθεί αυτό με τον οικονομικό συντονισμό, διότι δεν είναι αμυγό θέμα κρατών μελών αυτό. Θα πρέπει να ορίσουμε την ανάπτυξη, την οικονομική, ε, για να έχουμε μια καλή δημοσιονομική στρατηγική θα πρέπει να έχουμε και μια στρατηγική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Αλλιώς πολύ δύσκολα θα ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Για την ανταγωνιστικότητα δεν είναι θέμα κάθε χώρας ξεχωριστά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε μια σύγκληση με στόχους παγκόσμιους. Σύγκληση λοιπόν της ανταγωνιστικότητας χρειαζόμαστε και μεγαλύτερο συντονισμό. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για το νομισματικό και δημοσιονομικό συντονισμό. Είπαμε, ο οικονομικός συντονισμός έχει δύο σκέλη. Εσείς κάνετε νομισματική πολιτική, η οποία συνεισφέρει ε, στη ρευστότητα και στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η νομισματική πολιτική, κατά με, είναι κάτι ε, το οποίο οδηγεί σε διακρίσεις. Δηλαδή όπου έχουμε προβλήματα τα λύνουμε και δεν έχουμε ενιαία προσέγγιση προς όλους. Δεν κάνουμε το ίδιο με τη δημοσιονομική πολιτική. Η νομισματική αντιμετωπίζει ε, κάθε φορά ένα πρόβλημα με προσαρμογή χωρίς να αντιμετωπίζει το σύνολο. Πάλι δεν έχουμε συντονισμό εκεί. Όσον αφορά την ε, νομισματική πολιτική, κοιτάξτε, η εντολή μας είναι σαφή. Σταθερότητα των ε, ε, τιμών σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων και σε 16 χώρες. Τι έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω το μέσο ετήσιο πληθωρισμό τα τελευταία 11,5 χρόνια φτάνω στο αριθμητικό στοιχείο του 1,98%. Πολύ ακριβές. 1,98% σε 11,5 χρόνια μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην ε, Ευρωζώνη από τότε που άρχισε να λειτουργεί. Πρέπει να πω λοιπόν ότι συνάδει πλήρω ε, με τον ορισμό μας ε, της ε, σταθερότητας των τιμών κάτω από το 2% και είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια τέτοια χρονική περίοδο για χώρες και κεντρικές τράπεζες που ήταν οι γονείς, για να το πω έτσι, της Ευρωζώνης. Οπότε, Σύμφωνα με τις ε, προβλέψεις μας, φέτος, το τέλος του έτους, θα είμαστε για μία δωδεκαετή περίοδο στο 1,96 ή 1,97% θα δούμε τι θα γίνει ανάλογα με τον ανταγωνισμό και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μας ε, καθήκον. Οι συμπολίτε μας γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται σε εμά ε, για να ε, επιτύχουμε τη σταθερότητα των τιμών μέσω πρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όπως βλέπετε μίλησα για μια δωδεκαετή περίοδο. Το κάνουμε αυτό ό,τι κι αν γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα τη ε, εντολή του καθήκοντο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είτε οι δημοσιονομικέ πολιτικέ είναι εξαιρετικέ, είτε όχι. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη ζωή μα το να είναι εξαιρετικές, ε, γιατί δεν υπάρχει, πληθωριστικό, δεν υπάρχει το στοιχείο του πληθωρισμού στι καλέ δημοσιονομικές πολιτικέ. αλλά και στην περίπτωση των κακών δημοσιονομικών πολιτικών, όπω ισχύει αυτή τη στιγμή, κάποιοι τα καταφέρουν καλύτερα από άλλου, αλλά έχουμε κάποιε δυσκολίε. Πρέπει όμω να επιτύχουμε τη σταθερότητα των τιμών και πρέπει να είμαστε και αξιόπιστοι ω προ τη σταθερότητα των τιμών. Πρέπει να πείσουμε του παρατηρητέ, του συμπολίτε μα, τι επιχειρήσει και τους ότι κατά τα ερχόμενα έτη θα εξακολουθήσουμε να έχουμε σταθερότητα των τιμών, κάτι που πρέπει να πω ισχύει. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, οι πληθωριστικές ε, προσδοκίες συνάδουν ε, με τον ορισμό μας της σταθερότητας των τιμών για τα επόμενα έτη. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ε, βασικό ε, στοιχείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, δεν έχουμε μόνο πολύ καλό ιστορικό από τότε που υπάρχουμε, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να εγγυηθούμε και για το μέλλον επειδή αναφερθήκατε και στο συντονισμό, τα λέω όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας ανεξαρτήτως των συνθήκων και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ε, υπό συγκεκριμένε συνθήκες με πλήρη ανεξαρτησία τότε βεβαίω ε, δεν ε, θα μπορούμε να παραμείνουμε στις προβλέψεις πληθωρισμού που ανέφερα και δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την εμπιστοσύνη που και οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας αλλά και οι συμπολίτες μας οι ίδιοι περιμένουν από μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Σιλβή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτά τα οποία κάνατε τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί από τον καιρό που σας είδαμε τελευταία φορά έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δημοσίευσε μία έκθεση για την ε, διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Πολύ γεμάτο και πυκνό κείμενο. Εσείς πολλές φορές φαίνεται να είσαστε μόνος σας στην, ε, στην θέληση ε, να υιοθετούνται από κοινού οι αποφάσεις σε κάποιους τομείς, ε, όχι, να μην επιβάλλονται οι αποφάσεις από, την, από, την, από, από τις Βρυξέλλες όσον αφορά τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς, αλλά τέλος πάντων να υπάρχει κάτι, κάποια επιτροπή παρακολούθησης κτλ. ερωτώ με μήπως υποσκάθεται προστατεύεται με τον τρόπο αυτό η θέση της Κομισιόν και μήπως πολλοπλασιάζονται οι οργα... τα διάφορες επιτροπές, οργανισμοί κτλ. Διότι υπάρχει μια ε, διασπάθηση αν θέλετε των αρμοδιοτήτων και στο κάτω-κάτω θα πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η ευθύνη της Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι υπόλογη ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Οι επίτροποι μπορεί να έρθουν εδώ και μπορούν να ε, μας πούνε τι κάνουν. Και από την άλλη πλευρά το Κοινοβούλιο τι μπορεί να κάνει ε, για να ενισχύσει αυτή αν θέλετε την, ε, το συντονισμό σε θέματα τα οποία είναι κοινή αρμοδιότητες και στη συνεργασία και με τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Πολλά πράγματα όπως είπατε έγιναν από την τελευταία μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπατε. Στο σημείο 6 της ε, θέσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υπευλήθη και υποβλήθηκε στον πρόεδρο Βαν Ροπόη και δημοσιεύθηκε, αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία, η δημοσιονομική ανεξάρτητη υπηρεσία, η agency που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε μια σωστή διάγνωση ε, για τους προϋπολογισμούς των διαφόρων ε, κρατών της Ευρωζώνης αλλά και για να επιτρέψουμε ε, να έχουμε έναν συνεχή έλεγχο της μεσονικής κατάστασης των κρατών μελών, λέμε ότι θέλουμε να βρίσκεται στο εσωτερικό της Κομισιόν. Εμείς αυτό προτιμούμε. Επομένως, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό σε κάποιους τομείς υπάρχει η δυνατότητα στο εσωτερικό της Κομισιόν να, να υπάρχουν κάποιες μονάδες ή κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να είναι ανεξάρτητες, που μπορούν να είναι ανεξάρτητες, δηλαδή θα πρέπει να ε, εκμεταλλευτούμε ό,τι μας προσφέρει το παράγωγο δίκαιο και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι λέμε ρητά ότι δεν θέλουμε να θίξουμε τις αρμοδιότητες και τα προνόμια της Κομισιόν όσον αφορά ε, τις προειδοποιήσεις ή τις προτάσεις που υποβάλλει η Κομισιόν. Και στην εισαγωγική μου ομιλία είπα ότι σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, θέλουμε η Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να αντιστραφούν μόνο με, την, με ομοφωνία από πλευρά των κρατών μελών. Δηλαδή, επαναλαμβάνω και αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι σε αυτόν τον τομέα που όπως και εσείς είπατε είναι κρίσιμος και ζωτικής σημασίας, Θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο, ένα σύστημα επίβλεψης που να είναι σαφές και σταθερό, διότι η εμπειρία μας έδειξε ότι εκεί πάσχουμε, σε αυτόν τον τομέα πάσχουμε. Επομένως αυτή η ανεξάρτητη υπηρεσία στο εσωτερικό της Κομισιό ενδεχόμενα μας ικανοποιεί πλήρως. Μιλήσαμε για την Ελλάδα πριν από λίγο. Ε, προφανώς δεν μας επιτρέπεται να αντιμετωπίσουμε δεύτερη φορά τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή εννοώ να έχουμε μια σαφή και σωστή διάγνωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κυρία Τρισέ για τις παρατηρήσεις σας και επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά από την τελευταία φορά ε, που ήσασταν εδώ πριν από μερικούς μήνες ήταν λίγο δύσκολο να περιορίσουμε την ερώτηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά εν ώψη της ανακοίνωσης του Σαββάτου της Κινέζικης Κεντρικής Τράπεζας ε, ότι δεν θα είναι πια συνδεδεμένη με το δολάριο και συνεπώς ε, θα γίνει επανεκτίμηση ε, σε σχέση με το δολάριο του νομίσματός σας. Θα ήθελα να μας πείτε Πώς επηρεάζει αυτό τις προοπτικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν επηρεάζει τις τιμές, ε, τους δείκτες τιμών ε, ή αν δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως αν θα έχει αποτέλεσμα αυτό και στις χώρες εκτός Ευρωζώνης επειδή υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλες εισαγωγές αγαθών από την Κίνα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η απόφαση την οποία δημοσίευσαν οι κινέζικες αρχές Νομίζω ότι είναι μία καλή απόφαση που κατά την άποψή μας εξυπηρετεί την ίδια την Κίνα, την ανάπτυξη της Κίνας, την οικονομία της Κίνας και είναι επίσης προς όφελος ε, των εταίρων της Κίνας, δηλαδή της παγκόσμιας ε, ε, οικονομίας. Πηγαίνει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης σταθερότητας και μεγαλύτερης ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους τους εταίρους. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει όταν Είχαμε πάει στο Πεκίνο με τον κύριο Γιούνκερ, με τους ε, ε, αρμόδιους επιτρόπους ε, και είχα πάει κι εγώ. Πρέπει να πω λοιπόν ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η απόφαση αυτή και πιστεύω ότι είναι μια καλή απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ Λαμπέρς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Την τελευταία φορά που ήρθατε προσοχή στατικές εξόδου, όχι πολύ γρήγορα, όχι πολύ δυνατά. Τώρα σώζουν αυτό ο θήκον, πολιτικές λιτότητας. Λέτε δημοσιονομικά υπεύθυνα και βιώσιμα. Δεν διαφωνούμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγαίνει από το ρόλο της όταν υπαγορεύει πώς να φτάσουμε σε ισοσκελισμένο προπολογισμό και απλώς επιβάλλει περικοπές. Πάντω σωστά τα λέτε, σας ακολουθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ανησυχούμε η οικονομία δεν ξαναμπαίνει στις ράγες περικόπτοντας τις κοινωνικές βάσεις και ταυτόχρονα χωρίς να επενδύουμε στο μέλλον. Οι πολιτικές λιτότητας βεβαίως περιορίζουν τις δυνατότητες επενδύσεων. Και θέλετε μια δημοσιονομική ομοσπονδία, συμφωνούμε για την εποπτεία, για τις δαπάνες, αλλά λείπει ένα σημαντικό σκέλος εδώ και ποιο είναι αυτό, εποπτεία και των εσόδων, γιατί ορισμένοι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών ε, εμποδίζουν ε, και άλλες χώρες από κάποια έσοδα γιατί έχουμε εδώ ένα φορολογικό ανταγωνισμό. Και πού είναι λοιπόν αυτό το δεύτερο σκέλος της ε, Δημοσιονομικής Ομοσπονδίας. Χρειάζεται μεγαλύτερη φορολογική συνεργασία και μια που μιλάτε για αυτά τα θέματα θα ήθελα την άποψή σας. Και για μας Δημοσιονομική Ομοσπονδία σημαίνει πολιτική ομοσπονδία γιατί το υπαριθμό ένα ζήτημα σε κάθε χώρα κυρίαρχη είναι ο προπολογισμό της στην κατάσταση που βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των κρατών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, λέει ο κύριος Τρισέκη, όχι μόνο των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά γενικά των ε, βιομηχανικών κρατών στον κόσμο μας. Είναι σαφές ότι η προοπτική επιστροφής σε μια βιώσιμη κατάσταση καλής, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι εκ των ουκ άνευ και καθόλου αντιφατική με την ανάπτυξη. Αντίθετος, είναι απαραίτητη για να υπάρξει και ανάπτυξη, ε, να εδρεωθεί η ανάκαμψη της οικονομίας και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Για ποιο λόγο. Απλούστατα, διότι εάν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των κρατών να ανακτήσουν τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών τους, τότε τα νοικοκυριά δεν θα καταναλώνουν όσο θα έπρεπε και δεν θα επενδύουν από φόβο οι ίδιες επιχειρήσεις δεν θα προετοιμάζουν το μέλλον οι δε επενδυτές θα ξέρουν ότι θα έχουν ε, δυσκολίες να ε, πάρουν τα χρήματά τους πίσω και θα ζητούν μεγαλύτερα επιτόκια. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν. Το πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε δεν είναι απλώς ευρωπαϊκό. Και βεβαίως δεν είναι πρόβλημα της Ευρωζώνης και μόνο, αλλά όλων των βιομηχανικών κρατών στο σύνολό τους. Και όλες οι χώρες αυτές μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο σε αυτή τη στρατηγική ανάκτηση της εμπιστοσύνης και των καταναλωτών και των επενδυτών και των επιχειρήσεων. Και πάλι εδώ βλέπω συμπληρωματικότητα και καμία αντίθεση μεταξύ εδραίωσης της ανάκαμψης και δημοσιονομικής φρόνησης. Έρχομαι τώρα στην ε, φορολογική συνεργασία. Αυτό είναι ένα ευρύτατο πεδίο όπου ε, και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα. Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο οι δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η φορολογική συνεργασία και η φορολογική εναρμόνιση που μπορεί θεωρητικά ο καθένας να εύχεται δεν είναι δυνατή όσο θα επιθυμούσαμε. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες λοιπόν και ε, τη φορολογία και τα Γι' αυτό ακούτε συχνά να λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πολύ σημαντικές οικονομίες στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μόνο του θα οδηγήσει, θα βοηθήσει για τη φορολογική εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε φαίνεται ότι πολλά μέλη της Επιτροπής και η δική μας ε, Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, κατηγορούν τους οργανισμούς ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για το πώς βαθμολογούν τα, το δημόσιο χρέος. Και πραγματικά με δυσκολία αντιμετωπίζω τις απόψεις αυτές, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και τις δικές σας. Εδώ ασχολούμαστε με το θέμα τα αρχής βέβαια, έτσι. Εάν, εάν πάτε ας πούμε σε έναν αγώνα υπασίες ε, και ποντάρετε σε ένα άλογο το οποίο έρχεται τελευταίο ποιος θα φταίει εσείς ε, που, ποντά, ποντάρατε στο άλογο αυτό φταίει το άλογο φταίει ο, ο, ο αναβάτης ε, φταίνε αυτοί που, κάνουν, που βάζουν τα στοιχήματα ποιος φταίει τι να σας πω, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν στοιχηματίζω στις υποδρομίες. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πηγαίνω ούτε σε κανένα, ούτε Άρτου Τριόμφ ούτε σε κανένα άλλο αγώνα υπασίας ε, στον υπόδρομο γενικώ. Αλλά να σας πω ότι δεν φτάνουν να χαρτί οι οργανισμοί αξιολόγησης ε, ε, πιστοληπτικής ικανότητας αλλά γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της τελευταίας χρονιάς και μετά από όλα όσα είδαμε και το 2007, 2008 και 2009 και σήμερα, είναι ότι υπάρχει μια κυκλική εξέλιξη της οικονομίας, αν θέλετε, ε, και υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις που επηρεάζονται από τέτοιου είδους ανακοινώσεις διότι αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα. Αυτό δεν συμβαίνει όμως όταν δείτε τι συμβαίνει. Και δεν κατηγορώ κανένα, μια παρατήρηση κάνω που λίγο πολύ αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Όλοι θέλουμε σταθερότητα όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, αν θέλετε. Επομένως, κάποια στοιχεία, κάποια στοιχεία προωθούν, αν θέλετε, σε κάποια αστάθεια. Αυτό, αυτό είπα μόνο. Και οι G20 προσπαθούν ε, να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Και πραγματικά θα πρέπει να δούμε ε, πώς συνεισέφεραν στην κατάσταση αυτή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, αυτοί οι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και άλλοι παράγοντες γενικότερα. Και θα πρέπει ακριβώς ε, θα πρέπει να βρούμε πώς ε, μπορούμε όλοι αυτούς τους παράγοντες να τους κάνουμε να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε σταθερότητα. Ο κύριος Πόρτας ακόμα τον περιμένουμε μήπως να το αναβάλουμε λίγο. Θα έρθει ο κύριος Πόρτας, θα πρέπει να κάνει μόνο τη σύνοψη της έκθεσης του και έρχεται. Okay, that's, that, that, that's fine. Εντάξει. Ο κύριος Τόλογιαν. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, από δύο χρόνια, εδώ πάλι, στην Επιτροπή αυτή, Αναφέρατε ποιε ε, θα μπορούσαν να είναι οι μελλοντικέ τάσει ε, στις ε, πιέσει που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και έχετε δίκιο. Πράγματι έγινε αυτό και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ακρίβεια της ανάλυσης που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για τα κράτη της Ευρωζώνης, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, έχετε αυτό το πρόγραμμα ε, αγοράς κρατικών ομολόγων. Αν ένα κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης ε, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που σας οδηγούν στο να ε, έχετε αυτό το πρόγραμμα, θα κάνατε το ίδιο. Κοιτάξτε. Οι συστάσεις και οι προτάσεις ε, δεν είναι διάλεξη στις υπόλοιπες κεντρικές ε, τράπεζες και πολλοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψη όταν ε, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και είναι πολύ δύσκολη απόφαση όταν πρέπει να ληφθεί. Όπως βλέπετε, κάναμε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν, γιατί άλλες κεντρικές τράπεζες που είχαν προβεί σε αυτές τις αγορές ομολόγων, το είχαν κάνει αυτό ως τμήμα ε, ενός προγράμματος ε, που αφορούσε την ενίσχυση της ρευστότητας ε, στην οικονομία. Και δεν είναι αυτό ε, ίδιο με αυτό που κάναμε εμείς. Εμείς προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την αποκατάσταση μιας, ενός μηχανισμού ε, καλύτερης νομισματικής πολιτικής ε, σε επίπεδο ευρωζώνης. Και αυτό το λέω για να σας δείξω ακριβώς ότι πρέπει πάντοτε να ε, βλέπει κανείς την ιδιαιτερότητα της κατάστασης και γι' αυτό δεν θα έκανα ε, τέτοιου είδους συστάσεις σαν αυτές που με ρωτήσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λούλινγκ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, αν είχα χρόνο, θα σας έκανα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα σχόλιά σας που δημοσιεύτηκαν στη σημερινή Λιμπερασιό ως προς τη συμπεριφορά του επικεφαλής της Bundesbank. Και είχε την αυθάδεια, το άκρο άτο της ε, αλαζονίας να φιλοδοξεί να σας αντικαταστήσει. Συγχαρητήρια για τα όσα απαντήσατε και σε ό,τι αφορά τον τυχοδιοκτισμό σας. Υποτιθέμενο. Έρχομαι στην ερώτησή μου. Δηλώσατε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται δημοσιονομική ομοσπονδία. Και επαναλαμβάνω τα λόγια σας και παραθέτω για να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρή. Αυτό θα πρέπει να αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των δημοσίων οικονομικών και των πολιτικών τους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς χρησιμοποιείται αυτό το στοιχείο στη συζήτηση που γίνεται για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τις προόδους προς την οικονομική διακυβέρνηση γίνονται νέες συζητήσεις θεσμικού χαρακτήρα. Ορισμένα κράτη, μεταξύ αυτών ε, ένα που γνωρίζετε όλος ιδιαιτέρως, ζητούν ε, να κυριαρχήσει η διακυβερνητική λογική και διάσταση. Δεν το θεωρείτε αυτό περίεργο. Κάποιος το ανέφερε, δεν θα έπρεπε να ενισχυθεί μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη συνήθεια να δίνουν αμνηστία στον εαυτό τους. Θα γνωρίζετε καλά αυτά. Ε, τα γεγονότα των τελευταίων ετών είναι πάρα πολύ εύγλωτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ε, σε ό,τι αφορά τη Δημοσιονομική Ομοσπονδία. Εγώ σας είπα ότι χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο με μια ομοσπονδία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολιτική ομοσπονδία η Ευρώπη. Έχουμε ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν είναι πολιτική ομοσπονδία η Ευρώπη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κανόνες υπερβολικά σοβαρούς για την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών. Αυτό ε, χαρακτηρίζω εγώ ε, ως αντίστοιχο με την οικονομική δημοσιονομική ομοσπονδία που δεν υφίσταται. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών συγγνώμη, και της ανταγωνιστικότητας. Και εντός της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή ε, τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και την παραγωγή. Αυτό σας είπα, αυτό ε, φρονούμε και μιλώ και εξ ονόματος ε, του Συμβουλίου Δίκτων ότι θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ ουσιαστικά να έχουμε ένα ποιοτικό άλμα στην εποπτεία αυτών των πολιτικών και των δημοσιονομικών αλλά και της ανταγωνιστικότητας. Όπως σας είπα προηγουμένως θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε ε, τις δυνατότητες που μας δίνει το παράγωγο δίκαιο. Γιατί δεν είναι ούτε πάρα πολύ εύκολο, ούτε πάρα πολύ ε, γρήγορο ε, το ενδεχόμενο και η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της συνθήκης. Η διακυβερνητική λογική την οποία αναφέρατε, τι είναι. Συνδυασμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέραμε την Επιτροπή και το πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει και του Συμβουλίου, το οποίο και το Συμβούλιο έχει και αυτό το ρόλο του να παίξει. Αλλά δεν είμαστε σε μια διακυβερνητική λογική. θα πρέπει να είμαστε εκεί στην καρδιά της κοινοτική μεθόδου, όπως την αντιλαμβανόμαστε και ισχύει από την αρχή της ίδρυσης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχει να διαδραματίσει ρόλο και, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η εποπτεία και ο έλεγχος μεταξύ ίσων, το peer review. Ε, το πρώτο δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάσα καθόλου, να διαβάσετε τι είπα εγώ και τι απάντησα. Ουδέν σχόλια. Εκτός μικροφώνου, κυρία Λούλη, δυστυχώς. Ε, Η Κόριν Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, κύριε Πρόεδρε Τρισέ, θα ήθελα να σας επενέσω για το στιβαρό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε ε, και διευθύνεται ε, τις καταστάσεις και τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Μιλάτε για ενίσχυση της κοινοτική μεθόδου και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Συμφωνώ απολύτως. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για κάτι άλλο. Είπατε ότι η αύξηση των δανείων προς τι επιχειρήσεις είναι αρνητική ακόμα. Γιατί πραγματικά οι επιχειρήσεις χρειάζονται το κεφάλαιο τώρα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όμως την περασμένη περίοδο επιλέξατε να δώσετε πολλά χρήματα για να ενισχύσετε σχεδόν δωρεάν τη ρευστότητα των τραπεζών, ε, αλλά ε, οι τράπεζες επενδύουν σε κρατικά ομόλογα, σε κρατικά ε, δάνεια. Και τώρα μιλάμε για το τεστ αντοχής. Τι γίνεται με τις τράπεζες που έχουν χαμηλή ρευστότητα. Θα κάνετε και άλλη ένεση ρευστότητας προς τις τράπεζες. και αν επενδύσουν και πάλι σε κρατικά ομόλογα αντί να δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις, τι θα γίνει. Πού θα βρουν το κεφάλαιο οι επιχειρήσεις. Τι μέσα και τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ε, αν ε, αποδειχθεί και πάλι ότι πάσχουν από ρευστότητα οι τράπεζες. Thank uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς ε, όσον αφορά τα δάνεια ε, που βρίσκονται σε κρεμότητα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο προτείνουμε τώρα είναι να έχουμε ένα ε, εργαλείο, αν θέλετε, για τα εκρεμή δάνεια που ε, θα έχει δύο στοιχεία, ένα αρνητικό και ένα θετικό κυρίως καταρχάς όσον αφορά τα δάνεια στα νοικοκυριά. Εκεί βλέπουμε ότι η ανάκαμψη της ανάπτυξης έρχεται πριν από την ε, ανάκαμψη στον ε, τομέα των επιχειρήσεων. Αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση. Επομένως έχουμε ένα 2,5% συν για τα, ε, για τα νοικοκυριά και μείον 2,6% μείον εκεί για τις επιχειρήσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται με αυτό το οποίο είχαμε διαπιστώσει στο παρελθόν σε παρόμοιες καταστάσεις. Περιμένουμε ότι προοδευτικά ο δυναμισμός των δανείων προς τις επιχειρήσεις να να προχωρήσει και να υπάρχει μια ανάκαμψη. Ε, τώρα βέβαια αυτό το οποίο ζητάμε από τις τράπεζες να κάνουν είναι να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις τράπεζες και το ξέρουν και τους το λέμε συνέχεια ότι αυτό το οποίο γίνεται από, την, ε, από τις κεντρικές τράπεζες ε, και δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή γενικότερα ε, την Ευρωζώνη, αλλά αναφέρομαι και στις άλλες κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης αλλά και του, των υπολείπων χωρών, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε νομισματικές πολιτικές μεν, με στάνταρ ή μη στάνταρ μέτρα, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο τον στέλνουμε συνεχώς και ε, θα πρέπει όλοι και οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να υιοθετούν μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία. Όπως ξέρετε τώρα, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτά τα τεστ κοπόσεως, τα, stress tests, θα δημοσιοποιούνται για όλες τις τράπεζες. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο και ζητάμε από όλους τους εταίρους μας, αν θέλετε, να ε, εργαστούν ε, και να είναι πολύ δραστήριοι, διότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να φροντίσουν να έχουμε την σωστή διάγνωση και την κατάλληλη ε, θεραπεία, εάν και εφόσον ε, χρειάζεται θεραπεία ε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ κοπόσεως. Όλα αυτά συντονίζονται ε, από μας και γίνονται σε επίπεδο 27 και συνεργαζόμαστε και με την Κομισιό. έτσι ώστε να γίνει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αυτή η άσκηση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική πρέπει να γίνει αυτό το τεστ κοπόσεως με, έναν ιδιαίτερο επαγγελματικό τρόπο για να στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λίον Βαν Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υποστηρίξω στην απόφαση που πήρατε να, να υιοθετήσετε κάποιες ρυθμίσεις για τις χώρες των οποίων, ε, που έχουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέος τους. Και ε, από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κινδύνους ε, πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι γύρω στο 1%. Δεν υπάρχει κίνδυνος επίσης να επηρεάσει ο πληθωρισμός, να επηρεαστεί μάλλον ο πληθωρισμός από το κόστος, διότι ούτως ή άλλως οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι. Τέλος πάντων, τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Ε, θέλετε να έχουμε μία ε, δημοσιονομική πολιτική η οποία να, δια, ε, να είναι ε, κάπως περιοριστική με βάση τις πολιτικές εξόδου. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως, ότι όχι μόνο οι επενδύσεις ε, ε, φαίνονται αδιάφορες όσον αφορά τα επιτόκια, αλλά τα επιτόκια δεν μειώνονται, διότι από ό,τι φαίνεται έχουμε πέσει σε μια παγίδα, αν θέλετε, ρευστότητας. Ε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, εφόσον τα κατάλληλα, τα βασικά, τα αρχικά χρέη δεν είναι τόσο καταστροφικά, το ελλείμματα, συγγνώμη, μήπως είναι κατάλληλο να πρεσβεύουμε μια πολιτική λιτότητα η οποία θα πλήξει την ανάκαμψη. Για το πρώτο θέμα που μου αναφέρατε, γιατί όπως είδατε και ακούσατε, εμείς ανακτούμε όλη τη ρευστότητα που δίνουμε στο πλαίσιο αγοράς ε, ομολόγων. Οπότε, το σύνολο της ρευτότητας το ξαναπαίρνουμε πίσω ευρώ προς ευρώ. Και όσον αφορά το δεύτερο θέμα που θίξατε, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι μόνο εντός της Ευρωζώνης, αλλά και εκτός ε, της Ευρωζώνης σε ε, βιομηχανισμένες χώρες, υπάρχει δυσπιστία και αυτό αντίκεται ε, στην ε, ε, εξυγίανση, γιατί αυτό δημιουργεί δυσπιστία και στους καταναλωτές και στους πολίτες, γιατί οι δημοσιονομικές πολιτικές που είναι περιοριστικές, εμείς θεωρούμε ότι ε, πρέπει να δημιουργούν εμπιστοσύνη στους ε, επενδυτές ώστε να μπορούμε και εμείς να επανέλθουμε σε μια βιώσιμη κατάσταση ε, μακροπρόθεσμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αν, ε, στις περιπτώσει βλέπουμε ότι αν δεν υπάρξει διόρθωση της κατάστασης, τότε μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να ανακάμψουμε και γι' αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες. Άρα, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των ε, πολιτικών που θα τις χαρακτήρισα σοφή, ε, πολιτικές σοφίας και επιστροφής σε μια κατάσταση βιώσιμη υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξηγήσατε λεπτομερώς και πλήρως νομίζω τους λόγους που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην απόφαση να αγοράζει εθνικά ομόλογα από την δευτερογενή αγορά και απαντήσατε με απόλυτη επάρκεια σε όλες τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στην απόφασή σας αυτή Πρόκειται ωστόσο για μια απόφαση προσωρινού χαρακτήρα. Είπατε πριν από λίγο είναι μια απόφαση περιορισμένης διάρκειας. Ήθελα να σας ρωτήσω ε, εάν μπορείτε να μας δώσετε κάποια ιδέα για το χρόνο διάρκειας αυτής της απόφασης και αν έχετε κάποιες σκέψεις για την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί μετά ε, εάν δηλαδή υποστηρίζετε την ιδέα δημιουργίας ενός ειδικού φορέα ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αγοράς εθνικών ομολόγων και έκδοσης ευρωομολόγων για παράδειγμα ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο κόστους δανεισμού για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. έχετε προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου θεσμού διαχείρισης κρίσεων με κεφαλαιακή επάρκεια. θα μπορούσε ίσως η επέμβαση στην δευτερογενή αγορά ομολόγων να περιλαμβάνεται στις, ε, στις αρμοδιότητες μιας τέτοιας αρχής. Σας ευχαριστώ. the Την πρώτη σας ερώτηση. Θα έλεγα ότι όπως συμβαίνει με όλα τα έκτακτα μέτρα, μη στάνταρτ, Ας πούμε η ρευστότητα που δίνουμε περιορισμένης διάρκεια είναι ε, σε συγκεκριμένο σταθερό επιτόκιο. Ξέρουμε ότι η κρίση ξεκίνησε τη μέση Σεπτεμβρίου του 2008 και, και ε, ορισμένα έκτακτα μέτρα, όχι στάνταρ μέτρα, αρχίζουν και μετά σταματούν όπως ας πούμε η συμφωνία με τη Federal Reserve, όπως το πρόγραμμα ε, αγοράς ε, μετοχών, όλα αυτά είναι μέτρα μη στάνταρτ και δεν είναι μόνιμης εφαρμογής. Είναι πάντα προσωρινά και μεταβατικά. Αυτό είναι σαφέστατο. Τώρα, μην με ρωτήσετε τίποτα παραπάνω σχετικά. Μιλώ μόνο για τον προσωρινό χαρακτήρα τους και τα χαρακτηριστικά του ακριβώς είναι περιορισμένης διάρκειας και όχι μακροπρόθεσμα. Τώρα, αναφερθήκατε, αν κατάλαβα καλά, σε ομόλογα ε, τα οποία θα μπορούσαμε ε, να χαρακτηρίσουμε ευρωομόλογα. Γνωρίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είμαστε υπέρ των ευρωομολόγων. Ε, ε κοινή ε, συμμετοχή των κρατών μελών. Δεν το θεωρούμε σκόπιμο στην παρούσα φάση. Γνωρίζω ότι ακούγονται τέτοιες φωνές που ζητούν ευρωομόλογα, αλλά αυτή δεν είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και βεβαίω παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι κάνουν οι Ευρωπαίοι και το πώς εγκρίνουν ε, αυτό το ειδικό όχημα τα διάφορα κοινοβούλια αλλά δεν είναι κοινή και ομοσπονδιακή εγγύηση. Τα όσα σήμερα γίνονται και υιοθετούνται ως πολιτικές χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή και παρατήρηση γιατί ε, θα είναι πολλά τα διδάγματα που θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε από το πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης που προτείνουμε κι εμείς. Και είναι ένα από τα τρία σημεία του Φαν Ρόμπο και της ομάδας εργασίας που εξετάζονται αυτόν τον καιρό, όπως είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, Η ομάδα εργασίας Φαρόμπαϊ έχει εξετάσει δύο στοιχεία, αλλά όχι ακόμα αυτό το πλαίσιο για τη διαχείριση τη κρίση. Ευχαριστώ. Είδα, ήρθε και ο κύριο ε, Πόρτας, αλλά πρώτα ε, ο Ραμόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Ντομινίκ Στράουσκαν είπε πριν από έξι μήνε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι απώλειε τραπεζικού τομέα μπορεί να μην έχουν ακόμη εμφανιστεί. Είπε συγκεκριμένα οι απώλειες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί και είναι κρυμμένες ε, στους ισολογισμούς των τραπεζών και ενδεχομένως ε, μπορεί να φτάσουν μέχρι το 50%. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο, ο κύριος είπε ε, ότι η κατάσταση αυτή είναι, είναι εντονότερη στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Και το δεύτερο ερώτημα είναι στην Ευρωζώνη οι Ισπανικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη ε, ε, αναγνωρίσει απώλειες. Ο εποπτικός φορέας της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας είπε πριν από τρεις μήνες ε, ότι η κατάσταση οι απώλειες ε, είναι 450 δισεκατομμύρια, δηλαδή 45% ε, του ισπανικού ΑΕΠ. Ο πρόεδρος ε, του επιμελητηρίου είπε ότι 35% του ποσού αυτού δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακτηθεί. Ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το πλαίσιο σε σχέση με το ε, πρόγραμμα διάσωσης ε, της Ισπανίας. Πιστεύετε ότι η ανακεφαλαιοποίηση και η διαφάνεια θα ήταν προτιμητέα σε σχέση με το ε, ταμείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που κατά τη γνώμη μου δεν είναι επαρκώς διαφανές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο σας ερώτημα, Δεν έχω ιδιαίτερο σχόλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές εκατέρωθεν του Ατλαντικού σε σχέση με τις απώλειες ε, ή την αποκάλυψη των απολειών. Είμαστε βέβαια δύο οικονομίες ε, διαφορετικού, με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Ε, γνωρίζετε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε περνά πολύ από τις εμπορικές τράπεζες συγγνώμη, στην Ευρώπη περνά από τι εμπορικέ τράπεζες, ε, στην ε, Αμερική περνά από τις άγορε και επομένως είναι πολύ διαφορετικά, διαφορετικοί διαφορετικές παράμετροι που ε, υπησέρχονται. Δεν υπάρχουν πιστεύω μεγάλες διαφορές εκατέρωθεν του Ατλαντικού συνεπώς. βέβαια, τούτου λεχθέντος πιστεύω ότι το τεστ ε, κοπόσεως που αποφάσισαν οι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι αυτό που κάνουν οι Ισπανικές αρχές, ε, δηλαδή να συμμετέχουν στο τεστ αυτό, στο αυτό κοπόσεως, ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και συνεπώς θα φανεί ότι ε, σε μερικές περιπτώσεις η κατάσταση είναι καλύτερη από αυτή που φαίνεται, αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μια κατάσταση που πρέπει να ε, επιληθεί και όταν χρειαζόμαστε ε, κατάλληλε λύσεις πρέπει να εξευρεθούν αυτές οι κατάλληλε λύσεις. Ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει θα κάνω. Καταρχάς, δεν κατάλαβα. Γενικώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τα ευρωομόλογα. Θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλο τέλος πάντων. Πραγματικά δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τι, γιατί υπάρχει αυτή η στάση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ θυμάμαι ότι τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ένα επιτόκιο αναφοράς 5% και μέχρι τον Οκτώβριο αρνείται να κατεβάσει το, το, επιτόκιο αυτό. Επομένως ε, θέλω κάποια επιχειρήματα και όχι μία απάντηση του είδους δεν αρμόζει κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Εάν τα ευρωομόλογα ε, τα εξέδιδε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι θα φανταστεί, ποια θα είναι η άποψή σα. Δεύτερη ερώτηση, ε, την οποία εξετάζει η ομάδα Van Rompuy για το τελευταίο μεγάλο πακέτο. Πρέπει να δούμε πώς θα παρακολουθούμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η, επιταγή εν λευκό εκ προημίου δεν μου αρέσει. Πριν από την απόφαση των, του... των Εθνικών Κοινοβουλίων θα γίνεται κάτι τέτοιο και αυτό συνάδει με τις συνθήκες. Ε, I hope Ελπίζω ότι κατανόησα πλήρως την δεύτερη ερώτηση σας αλλά δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος ότι την κατάλαβα. Τέλος πάντων, για την πρώτη σας ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι μία θέση που έχει η Ευρωπαϊκή Τριγράψη εδώ και καιρό. Δηλαδή, ότι η κατάλληλη λειτουργία του πλαισίου στηρίζεται στην ενδυνάμωση της επίβλεψης. Και πριν από τα διδάγματα της, ε, της τελευταίας κρίσης, ε, εφαρμόζουμε τον τρόπο αυτό το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για μας αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Απ' την άλλη πλευρά, οι διάφορες κυβερνήσεις είναι υπεύθυνε για τις υπογραφές τους, για τις πολιτικές, δημοσιονομικές πολιτικές τους απέναντι στις, στους επενδυτές τους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Αυτό το θεωρήσαμε ότι είναι κομμάτι του πλαισίου, κομμάτι του τρόπου με, το, με τον οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει όσο μπορούμε τέλο πάντων το σύμφωνο σταθερότητα. Διότι αυτό ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Όμω το πνεύμα και το γράμμα της, του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη δεν εφαρμόστηκε. Και αυτό πρέπει να το διασώσουμε. Αλλά τέλο πάντων για τα ευρωομόλογα έχουμε διαμορφώσει μια άποψη αυτή, την άποψη αυτή, ανεξάρτητα από το ποιο τα εκδίδει. Κάτω από εξαιρετικές συνθήκες η Ευρώπη είδατε ότι βρήκε έναν τρόπο να ε, βρει μια λύση τέλος πάντων. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, φαίνεται ότι απευθυνόταν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ίσως να μην είμαι σίγουρος γιατί κατάλαβα. Τέλος πάντων, εάν θέλουμε να υπάρχει αλληλεξάρτηση που στηρίζεται ακριβώς στην ύπαρξη του ενιαίου νομίσματος, αν αυτή την αλληλεξάρτηση θέλουμε να την πάρουμε υπόψη μας, τότε θα πρέπει, ότι, θα πρέπει οι διάφορες δημοσιονομικές πολιτικές να, εξετάζονται από έναν ανεξάρτητο, από μια ανεξάρτητο, ανεξάρτητο οργανισμό, να αξιολογούνται από την Κομισιό και να εγκρίνονται από τους ομότιμους. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε αυτές τις εξαρτήσεις, αν θέλετε, που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σκληρό το μάθημα το οποίο λαμβάνουμε τώρα. Ότι ακριβώς πρέπει να υποστούμε, αν θέλετε, όλε τι συνέπειες ενό ενιαίου νομίσματο. Μοιραζόμαστε ένα κοινό πεπρωμένο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ο Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω αυτή τη στιγμή δεν έχω την αίσθηση ότι μας λείπουν εμπειρογνώμονες. Ε, μπορούν να καταρτήσουν, να μαγειρέψουν ε, προϋπολογισμούς. Αλλά υπάρχει το εξή βασικό σφάλμα. Ένα πολιτικό όργανο, οι Υπουργοί Οικονομικών, εκ των υστέρων επιπλέον, έρχονται να πούνε αν πήγαν όλα καλά. Αν φτάσαμε στο 3%, αλλιώς να λάβουν διάφορα μέτρα, γνωρίζοντας ότι καμιά φορά μπορεί να έρθει και δική τους η σειρά. Και όταν ο αμαρτωλός θα πρέπει να αποφασίζει για την τιμωρία, ε, θα είναι πολύ επίοικης με τους άλλους. Τι είναι αυτό το peer να τα κοιτάξουν εμπειρογνώμονες, δεν ξέρω αν είναι καλό. Και ε, ρωτώ, μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως είναι υπερβολικά πολιτική, πολιτικοποιημένη και την επηρεάζουν υπερβολικά οι διάφορες πρωτεύουσε των χωρών μελών με τις προτάσεις που κυκλοφορούν. Και ρωτώ, έχουμε ένα θεσμικό όργανο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αν κατάλαβα καλά τη συνθήκη είναι λέει και ανεξάρτητη. Και δεν ε, δέχεται υποδείξεις και... Ε, εντολές. Είναι η θητεία τους ε, άπαξ, μία θητεία μόνο και δεν μπορούν να τους πιέσουν για ανανέωση. Λοιπόν, αφού είναι λοιπόν ανεξάρτητο όργανο και ουδέτερο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μήπως θα πρέπει να διαδραματίσει κανένα πιο σοβαρότερο ρόλο και αφήστε τις γνωματεύσεις τους ειδικού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι και αυτή πολιτικά ελεγχόμενη. Εσείς ποιο ρόλο φαντάζεστε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, αυτό που είπατε για την ανάγκη να δρούμε εκ των προτέρων είναι κατά την άποψή μου βεβαίως ε, απολύτως απαραίτητο. Δεν μπορούμε μόνο εκ των υστέρων να κοιτάζουμε τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή έχουν ληφθεί γιατί δεν μπορούμε να ε, εργαζόμαστε σωστά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό. Στην πρόληψη, ε, να υπάρχει ένας αυτοματισμός αρκετά νωρίς στην κατάρτιση των προϋπολογισμών και στην εκτέλεση μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, πολύ πριν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατοφλιού 3% ή κάτι άλλο, να το παίρνουμε είδηση, να βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουμε προς την εκπλήρωση των πρόθεσμων στόχων. Να υπάρχει αυτόματη προειδοποίηση και αυτόματες κυρώσει αρκετά νωρί Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται ε, τις δυνατότητες που μας δίνει το παράγωγο δίκαιο. Αλλά επαναλαμβάνω, κατόπιν εορτής τι να το κάνουμε, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως, του λεχθέντος θα πρέπει να έχουμε εξίσου αυτόματες κυρώσει ή επιπτώσεις όταν ε, περάσει κάποιος αυτό το κατόφλιο 3% φερρυπίν. Στο παρελθόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τώρα, εμείς ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι είμαστε τμήμα της διαδικασίας. Και όπως γνωρίζετε, δραστηριοποιούμαστε και στο Eurogroup ε, και στο ΕΦΣΥ και σε ε, όλες τις ομάδες εργασίας. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, είμαστε διαθέσιμοι, είμαστε έτοιμοι. Τώρα έχει προκύψει ένα νέο συνδυασμό, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, σε σύνδεση, in liaison το λένε αυτό. Ε, άρα είμαστε πρόθυμοι να συνεργαζόμαστε και για να είμαστε ξεκάθαροι και με τους προσανατολισμούς μας σε ό,τι αφορά αυτό το ανεξάρτητο όργανο που θα ελέγχει και θα παρακολουθεί και θα υποπτεύει τις δημοσιονομικές πολιτικές, είπαμε ότι το προτιμότερο θα ήταν να βρίσκεται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ως ανεξάρτητος φορέας, παρότι είναι στην Επιτροπή. Ε, Κύριε Σμπάλτς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Ο Διεθνής Σύνδεσμος ε, Τραπεζών ε, συνήλθε στη Βιέννη και από ό,τι κατάλαβα εγώ χτύπησε τον κόδωνα κινδύνου ότι ε, όσο γίνεται ε, περισσότερες ρυθμίσεις ε, διακυβεύονται θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης. Μέχρι 10 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης σε ΙΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Είτε θα αποδομηθούν είτε δεν θα δημιουργηθούν. Αυτά όλα τι είναι, απλώς κινδυνολογία ή έχει δίκιο ο Διεθνής Σύνδεσμος των Τραπεζών. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση για τη βαθμολόγηση, την αξιολόγηση κρατών ολοκλήρων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι παγκοσμίω το καλύτερο όργανο για να αξιολογεί την ε, πιστοληπτική ικανότητα μελών, κρατών. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Δεν μπορείτε να γίνεται ένας οργανισμός τέτοιος αξιολόγησης για κράτη, επαναλαμβάνω. Και τρίτον, για το διατραπεζικό εμπόριο, ακούμε διάφορα να κυκλοφορούν, πολλά ερωτηματικά, πολλές απορίες. Αυτή τη στιγμή πώς αξιολογείται τη διατραπεζική αγορά στην Ευρώπη. Υπάρχει σταθερότητα, έχει ανακτηθεί, έχει αποκατασταθεί. <laughs> Όλα τα θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μου φαίνεται. Κύριε Χοντή. Θέλω να κάνω ερώτηση μετά, αν υπάρχει <laughs> Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία βασική εντολή που είναι πολύ σημαντική και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε σταθερότητα τιμών και δεν ξεχνούμε ποτέ ότι αυτός είναι ε, ο βασικός ε, γνώμονάς μας. Αλλά για τα υπόλοιπα ερωτήματά σας, θα ήθελα να πω ότι βλέπω συχνά στην ε, κοινότητα των εμπορικών τραπεζών υπάρχει συχνά αυτή η αίσθηση ότι οι κανόνες ε, τους οποίους επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Βασιλείας 3 ή στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της ομάδας των 20 ε, ή της Επιτροπής της Βασιλείας. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες ότι μπορεί να παρεμποδιστεί η ανάκαμψη. Και αυτό που απαντούμε είναι το εξής. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι μεσοπρόθεσμα ε, πρέπει να έχουμε έναν τραπεζικό τομέα που να είναι πολύ πιο ανθεκτικός. Πρέπει να εξηγήσουμε στις τράπεζες ότι αυτά που συνέβησαν στο 2008 και στο 2009, το 2008 και το 2009 ήταν πραγματικά τεράστια βήματα. Ο κίνδυνος ε, για το φορολογούμενο ε, εκατέρωθεν του Ατλαντικού τώρα είναι 27% του ΑΕΠ. Το γεγονός ότι είναι περίπου το ίδιο ποσοστό εκατέρωθεν του Ατλαντικού σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο βρισκόμασταν σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Δεν ε, το είχαμε καταλάβει αυτό. εμείς δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε αυτό. Συνέβη μία φορά για να αποφευχθεί μία τεράστια οικονομική ύφεση που θα ήταν πραγματικά δραματική. Υπήρχε ύφεση η οποία ήταν ήδη αρκετά σοβαρή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση και οι τράπεζες πρέπει να το κατανοήσουν αυτό. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του μόνιμου καθεστώτος ε, και ε, της ε, μεταβατικής κατάστασης. Πρέπει να δούμε τους κανόνες, τους κανονισμούς Μία σταθερή ε, κατάσταση για να εξασφαλίσουμε ότι, πρέπει να είναι, ότι θα είναι πιο ανθεκτικό το σύστημα για να μην υπάρχουν επιπλέον προβλήματα ε, στην πορεία προ την ανάκαμψη. Αυτό θα απαντούσα στην πρώτη σα ερώτηση. Στη δεύτερη ερώτηση δεν ε, βλέπω καμία εύκολη λύση ή σίγουρη λύση για το θέμα των ε, οργανισμών ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Έχουμε ήδη ένα σύστημα για να είμαστε να κάνουμε εκτιμήσεις προκυκλικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να πω. Και για το τρίτο θέμα που θέσατε, οι πιέσεις, οι, οι, εντάσεις μεταξύ των τραπεζών ήταν ένας λόγος ενεργοποίησης των μη συμβατικών μέτρων που έχουμε ε, λάβει στο παρελθόν και ελπίζουμε όλες οι αποφάσεις που ε, λάβαμε και οι νέες αποφάσεις ε, θα ενισχύσουν ε, σταδιακή επιτρο... στην ε, σταδιακή ε, επιστροφή σε μια ομαλότερη λειτουργία των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Τρισέ, τα προβλήματα των κρατικών χρεών είναι παρόντα και θα πρέπει να μας απασχολήσουν Μέχρι πριν από λίγα χρόνια σεβόμαστε τις, ε, τα όρια τα οποία επέβαλαν οι συνθήκες. Βέβαια υπάρχει μια γενική επιταγή που λέει ότι τα χρέη των κρατών μελών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 60% του ΑΕΠ. Φέτος η πρόβληψη είναι για 80% του ΑΕΠ. Όπως ξέρετε, επί του παρόντος ε, η πιο δραματική κατάσταση είναι η ελληνική. Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης πήραν αποφάσεις για να χρηματοδοτήσουν, να υποστηρίξουν την Ελλάδα και να σώσουν το γιούρο. Η λογική, η κοινή λογική που επικρατεί ανάμεσα στους πολίτες μας λέει ότι ναι, εντάξει, ε, τι κάνουμε τώρα. Οι πολίτες μέχρι τώρα ε, έσωζαν τις τράπεζες, τώρα θα σώσουν ε, και τις χώρες. Ποια είναι η απάντηση δική σας, η απάντηση του ανθρώπου που έχει γνώση στις ε, απανοτές ερωτήσεις που κάνουν οι πολίτες της Ευρώπης, που κάνει ο άνθρωπος, ο κοινός άνθρωπος. Ποιες θα είναι οι συνέπειες κατά την άποψή σας πάντα, αν η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρωζώνη για κάποιο χρονικό διάστημα και επανερχόταν όταν λύσει τα προβλήματά της και τα προβλήματα του υπερβολικού χρέους. Ποια θα ήταν η κατάσταση για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη. Επί του παρόντος, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της ιδέας. Όμως, ακούω συνέχεια τέτοιου είδους ερωτήσεις από πλευρά των συμπολιτών μου. Thank you very much. First of all... Καταρχάς, άκουσα αυτά που είπατε για τους 27 και το ε, χρέος τους ως προς το ΑΕΠ συμφωνώ απολύτως. Όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά μας παντού, σε όλες τις βιομηχανικές χώρες. Δεν είναι απορία άξιο που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη τον 27. Αν παίρναμε το G7 για παράδειγμα, θα βλέπαμε ότι το ετήσιο έλλειμμα ως κλάσμα του ΑΕΠ για τους περισσότερους από την ομάδα το 7 είναι 10, 10 και μισό 11%. η Ευρώπη ως σύνολο είναι κάτω ε, από αυτό το ποσοστό και η ίδια η Ευρωζώνη ακόμα. Το ετήσιο έλλειμμα αναθρηστεί φτάνει στο 6,5 με 7% του ελλείμματος, ετήσιο μιλώ. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι βιομηχανικές χώρες. Τώρα, για τη δεύτερη ερώτησή σας. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι πρόβλημα θα δημιουργεί το, αλλά για μένα αυτό δεν είναι καν υπόθεση εργασίας. Δεν θα επεκταθώ καθόλου σε αυτό. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Ιβο Στρίτζεκ. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου για τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσατε τα προβλήματα των κρατικών ομολόγων εδώ. Ξέρετε πολύ καλά βέβαια ότι πρόκειται για ένα βήμα καινούριο ε, που δεν έχει προηγούμενο που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ε, να παίρνει ομόλογα, κρατικά ομόλογα από την, την Ευρωζώνη. Θα μπορούσατε ίσως να μας εξηγήσετε γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες αυτών των αγορών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκάλυψε πληροφορίες ε, για ε, ποια κρατικά ομόλογα, ποιας χώρας ε, και πόσης διάρκειας ε, ήταν αυτά τα ομόλογα ή κατά ποιε συνθήκε συνθήκες ε, αγοράστηκαν τα ομόλογα αυτά. Ευχαριστώ. Εξήγησα τι κάναμε και γιατί αυτό το οποίο κάναμε είναι διαφορετικό από αυτά το, που, το οποίο γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιαπωνία, όπου υπάρχουν τέτοιου είδους αγορές με βάση του κατά πόσο είναι ποσοτικά εύκολο. Τώρα εμείς το κάνουμε για άλλους λόγους. Τέλος πάντων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει κάποιες πληροφορίες που αφορούν το ποσό, αν θέλετε, την ποσότητα αγοράς. Και το ποσοστό απόσυρσης τη ρευστότητα, έτσι ώστε να έχετε ένα, μια ιδέα για το τάξη μεγέθους. Ε, την πρώτη εβδομάδα είχαμε μια τάξη μεγέθου αγορών 16,5 δις, τη δεύτερη εβδομάδα 10 περίπου, την τρίτη εβδομάδα 8,5, την επόμενη εβδομάδα 5,5, μετά 6,5 και την τελευταία πληροφορία που έχω και που δόθη χτες, όχι σήμερα, σήμερα, είναι τέσσερα. Αυτό είναι το... Αυτή είναι αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε επί του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην δώσει παραπάνω πληροφορίες. Και αυτό, αυτό είναι το, αυτή είναι η τάξη μεγέθους και όσον αφορά τις αγορές και όσον αφορά την απόσυρση ρευστότητας από τις αγοράς. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ ένα ερώτημα και μετά ο κύριος Κουντής ε, είπε ότι και εκείνος θέλει να ρωτήσει κάτι, ενδεχομένως να έχουμε χρόνο και για έναν ακόμη ε, συνάδελφο. Κύριε Τρισέ, όταν ε, στην ομιλία σας αναφέρθηκατε στους ε, ισολογισμούς ε, που είναι ένας από τους ε, τρεις παράγοντες που ενίσχυσαν την παρέμβαση για την αγορά ελληνικών ομολόγων Βάση της οδηγίας για τις απαιτήσεις κεφαλαίων είναι μεγάλος ο δεν, δεν, δεν υπήρχε ονομαστικός κίνδυνος ε, για το νόμισμα αν ε, δεν μπορεί κανείς ε, δηλαδή να κάνει το... να τυπώσει το δικό του νόμισμα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν δυνατό αυτό χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταλαβαίνουμε τον κύκλο βέβαια στον οποίο έχετε βρεθεί τώρα και γι' αυτό ε, καταλαβαίνουμε την, ε, επικίνδυνη, τα επικίνδυνα αυτά μέτρα που λάβατε. Αλλά αυτή, αυτός ο αυτοματισμός για τον οποίο μιλήσατε, πώς θα ε, υπάρχει όταν ο κίνδυνος έχει άμεση σχέση με το χρέος των κρατών μελών και τι θα γίνει αν κάθε φορά πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει προβλήματα ελλημάτων των ε, κρατών ε, ε, μελών γιατί αυτό αυτομάτως θα είχε αντίκτυπο στη στάθμιση του κινδύνου, όπως επίσης και με την επιθυμία των ε, τραπεζών ε, να βοηθήσουν. Κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι σταδιακά μπορεί να ε, τις ξεφορτωθούμε αν η στάθμιση του κινδύνου δεν είναι επαρκής. Μήπως μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που με ρωτήσατε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και πρέπει να μελετηθεί. Είναι γεγονός ότι στο σύστημα αυτή τη στιγμή υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και αυτό είναι κάτι που είναι τμήμα της συζήτησης που κάναμε, της ευρύτερης συζήτησης και είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να ε, συντονιστεί σε περίπτωση που έχουμε ένα κοινό νόμισμα για πολλά κυρίαρχα κράτη. Το, ο βασικός λόγος για τον οποίο πάντοτε ε, θέλαμε τόσο πολύ να ε, γίνεται απολύτως σεβαστό και να εφαρμόζεται πλήρως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί όλα όσα είπατε έγιναν μετά την παρέκκληση από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. όλοι αποφασίσαμε, ήταν τμήμα της ε, συνθήκης του Μάστριχτ ε, και στην δευτερεύουσα νομοθεσία, ε, είναι κάτι το οποίο είναι... Δεν, δεν είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να μελετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή η συνάντηση με τον κύριο Τρισέ είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές, θα ήθελα υπό τη μορφή απολογισμού να τον ξαναρωτήσω δύο πράγματα που ρωτούσα όλο τον χειμώνα ε, και ομολογώ ο κάθε αρμόδιο και ομολογώ ότι ο κύριος Τρισέ έδινε κάποιες απαντήσεις. Επανέρχομαι λοιπόν κύριε Τρισέ. Τι επέβαλε και με ποιους όρους έχει μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη. Ποιος, ποιοι οι λόγοι που το φέρατε στην Ευρωζώνη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αισθανόσαστε σήμερα εσείς ανεξάρτητος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθώς από ό,τι διαβάζουμε στον τύπο στέλνει επιστολές σε εσά στην Κομισιόν υπαγορεύοντας και αυτό εποπτείες και κυρώσεις. Και η δεύτερη ερώτηση. Έχετε ξανασκεφτεί ανάμεσα στα διάφορα όπως είπατε σωστά λάθος θα εκτιμηθούν ποιοτικά άλματα, κβαντικά άλματα που πρέπει να γίνουν στην Νομισματική Οικονομική Ένωση μήπως πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως αποδείχθηκε τροποποιήστε σύμφωνα με τον παράγωγο δίκαιο όπως είπατε και αν το κατάλαβα καλά τη μορφή δανεισμού. Σας ρωτώ λοιπόν μήπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταλαβαίνουν τη δυσκολία χρειάζεται και αυτή ένα κβαντικό άλμα προκειμένου να παίξει καλύτερα το ρόλο της στην πρώτη σας ερώτηση. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξή μόνο. Στην περίπτωση της Ελλάδας είχαμε ένα ενιαίο πρόγραμμα που συζητήσαμε και αποφασίσαμε και έχει αποφασίσει μάλλον η ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φενός και, με τη, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρακολουθήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αποφάσισαν τελικά οι κυβερνήσει. Έχουμε λοιπόν ε, μία απόδειξη αυτού που θα χαρακτηρίζα καλή συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Φενό και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων αφετέρου. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτηση σα τώρα, θα έλεγα και πάλι το εξή. η βασική μας εντολή που απορρέει από τη συνθήκη και αυτό που ζητούν από εμά οι συμπολίτε μα είναι να εγγυόμεθα τη σταθερότητα των τιμών. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να είναι εγγυημένη η σταθερότητα των τιμών. Όταν είναι έκτακτε δε οι περιστάσει και όταν βλέπουμε ότι ούτε οι χρηματαγορέ ε, λειτουργούν ε, καλά, ε, όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία για κάποιο λόγο, η συγκεκριμένη χρηματαγορά, η ε, τάδε, η δίνα αγορά, όπως δυστυχώς διαπιστώσαμε πρόσφατα, που είχαμε και κραδασμούς και πάρα πολύ... Ε, μεγάλη ένταση της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης πρόσφατα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε τέτοια φαινόμενα, εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να ε, επανέλθει μια πιο φυσιολογική λειτουργία των αγορών. Αυτά χαρακτηρίζουμε αντισυμβατικά, μη συμβατικά μέτρα, not standard. Δεν εμποδίζουν κανονικά, ούτε πρόκειται ποτέ να εμποδίσουν το βασικό μας στόχο που είναι η σταθερότητα των τιμών. Και για το λόγο αυτό, όταν σας εξήγησα το πρόγραμμα για την αγορά ε, μετοχών, σας είπα ότι δεν αλλάζουμε ε, την νομισματική μας εντολή και παίρνουμε πίσω όλη τη ρευστότητα που είχαμε δώσει στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τρισέ. Νομίζω ότι εξαντλήσατε τις ερωτήσεις, ε, τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 27 στις 27 Σεπτεμβρίου, η επόμενη συνάντηση μαζί σας για το νομισματικό διάλογο, θα ήθελα να θυμίσω στα μέλη ότι είχαν προετοιμαστεί έγγραφα από τους εμπειρογνώμονες μας για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και πώς θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανείς τη συνθήκη για πιο ε, καλό συντονισμό